Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, να καλωσορίσω τους προσκεκλισμένους μας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ακρόαση για την μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής ε, και την πολιτική ε, διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων. Θα πρέπει καταρχάς να πω ότι εδώ είναι παρούσα η τηλεόραση του BBC η οποία θα μας ε, κινηματογραφήσει όλοι. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα. Ε, δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση. Ωραία. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους μας και νομίζω ότι σήμερα έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το ενδιαφέρον για αυτή την ακρόαση. Ε, έχουμε λίγους ευρωβουλευτές σήμερα εδώ, αλλά η Επιτροπή μας είναι μικρή και σήμερα δυστυχώς ε, συμπίπτει και με συνεδριάσεις άλλων επιτροπών. Ε, επομένως είναι δύσκολη παρουσία όλων εδώ. Να σας πω καταρχάς ότι η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής είναι για μας θέμα κεφαλιόδου σημασίας και εδώ στην Επιτροπή μας λέμε πάντα ότι η πολιτική διαχείριση και ε, διατήρησης των αποθεμάτων είναι η μόνη την οποία τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχουμε αγγίξει στις διάφορες μεταρρυθμίσεις της κοινή ελευτικής πολιτικής. Γι' αυτό και πολλοί από εμά θεωρούμε ότι είναι ο γόρδιος δεσμός ο οποίος χρειάζεται να τροποποιηθεί, εις βάθος μάλιστα, εάν θέλουμε η αλληλεία να έχει κάποιον μέλλον, κυρίως ε, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε και σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Χαιρόμαστε λοιπόν που ε, βρίσκεστε εδώ, άτομα εγνωσμένου κύρους, και να δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο τη ΦΑΟ, τον κύριο Βάλντι Μάρσον, ο οποίο είναι σύμβουλο του Γενικού Διευθυντή του Τμήματος ε, και Ιδατοκαλλιέργεια. Ε, πρόκειται για ένα άτομο πολύ γνωστό. Έχουμε λάβει πολλές φορές εκθέσεις που έχετε κάνει για τη θέση της ΦΑΟ για τα θέματα διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων. Γι' αυτό ακριβώς και μας ενδιέφερε όλους να σας προσκαλέσουμε εδώ για να μας εκθέσετε την ε, θέση της ΦΑΟ επί των θεμάτων αυτών. Έχετε το λόγο λοιπόν ε, για ένα τέταρτο κύριε Βαλτιμάρσον. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Γκρίμουρ Βάλτιμαρσον, είμαι από το τμήμα Αλλιάς και Δετοκαλλιέργειας του ΦΑΟ των Ηνωμένων Εθνών ε, στη Ρώμη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές που μου δίνουν τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για το ένα θέμα το οποίο με αγγίζει ιδιαίτερος. Όταν μεγάλωνα στην ε, χώρα μου, την Ισλανδία, το να είναι κάποιος αλλιάς ήταν κάτι το οποίο το έβλεπαν με πολύ θετικό μάτι οι αλείς ήταν αυτοί που έφεραν τροφή στο τραπέζι. Θεωρούνταν άνθρωποι γενναίοι και δυνατοί και κέρδιζαν ε, πάρα πολλά χρήματα. Εκείνη την εποχή η αλία ήταν ε, απλώς το να έχει κάποιος ένα σκάφος και να βγαίνει έξω στη θάλασσα να ψαρέψει. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο τομέας ε, παγκοσμίω πρέπει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ευτυχώς, ο λαός πλέον δέχεται ότι η αλληλεία δεν είναι απεριόριστη, τα αλλιεύματα δεν είναι απεριόριστα και θα πρέπει να υπάρχει ε, σημαντική διαχείριση. Η ΦΑΟ εργάζεται προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις επί του θέματος και έχουν εφαρμόσει πολύ σημαντικά ε, παγκόσμια μέσα για την παγκόσμια διαχείριση του Ισαλία και θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι σκέψει μα για το τι θεωρούμε χρηστή διαχείριση και τι είναι αυτό που κάνει τους αλληλείς να θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης των αλλιευμάτων. Θα πρέπει να ε, προσθέσω βέβαια αυτό που λέμε συνήθως, ότι οι απόψεις που αποτυπώνονται εδώ είναι οι δικές μου και δεν αντακατοπτρίζουν απαραίτητο στην άποψη της ΦΑΟ. Έχω μια σύντομη παρουσίαση, η οποία αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Καταρχάς θα σας δώσω μια, ε, ένα στιγμιότυπο της παγκόσμιας κατάστασης αλίας. Θα σα πω επίση γιατί οι αλληλεί δεν θεωρούν ότι η τρέχουσα διαχείριση των αποθεμάτων δεν είναι πολύ χρήσιμη. Θα σα πω επίση ε, ε, για του λόγου οι οποίοι κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να του ενθαρρύνουν να αλλάξουν άποψη και τέλο θα επισημάνω την συνεχή δέσμευση του, ε, της ΦΑΟ για να εφαρμόζει αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια και συστήματα διαχείρισή του που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην ευημερία, στην ασφάλεια των τροφίμων και στα βιώσιμα σχέδια για την κατανάλωση και την παραγωγή. Εδώ έχουμε τα στοιχεία. Η μπλε γραμμή δείχνει τα αλλιεύματα, η κόκκινη γραμμή είναι η υδατοκαλλιέργεια. Όπως βλέπετε, εδώ και δεκαετίες οι εκφορτώσεις αυξάνονται. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 σταμάτησε να αυξάνεται αυτή η τάση και περάσαμε στη στάσιμη φάση. Τα τελευταία 20 χρόνια οι εκφορτώσεις έφτασαν από τα ε, γύρω στα 82 με 84 εκατομμύρια τόνους για την ε, θαλάσσια αλληλεία και 10 εκατομμύρια τόνους για τις ε, ε ε, παράκτιες. Ε, συνεχώς έχουμε αύξηση και έχουμε και διπλάσια, ε, διψήφια αύξηση στην υδατοκαλλιέργεια, κυρίως στην υδατοκαλλιέργεια στην Κίνα. Προς ενημέρωσή σας, στο, αυτή τη στιγμή η υδατοκαλλιέργεια είναι το 44% όλων των αλλιευμάτων για που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αλληλεία μπορούμε να χαρακτηριστεί από τρεις φάσεις. Πρώτα είχαμε την ε, περίοδο του χρυσού πυρετού, αν θέλετε, όπου ε, θεωρούσαμε ότι ήταν ε, άπλετο το προϊόν και θεωρούσε κανείς ότι δεν υπήρχε καμία ανάγκη για περιορισμό. Αυτό φυσικά μας οδήγησε στην τρέχουσα κατάσταση της στασιμότητας που σας ανέφερα. Αυξήθηκε το κόστος και είχαμε και οικονομικές απώλειες ε, αλλά και απώλειες αλευμάτων. Και τώρα σε μια πρόσφατη έκθεση της ΦΑΟ και της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμούμε ότι ο τομέας αυτή τη στιγμή πετά από το παράθυρο περίπου 50 δις δολάρια ετησίως. Πάρα πολλά τα σκάφη, πάρα πολλά τα δίκτυα, πάρα πολλές ε, οι μηχανές και ούτω καθεξής. Τέλος, χρειαζόμαστε μία τρίτη φάση, μάλιστα τη χρειαζόμαστε απελπισμένα, είναι η περίοδος της αναγέννησης, έτσι την αποκαλούμε, και θα θέλουμε να έχουμε βιώσιμη, υπεύθυνη και οικονομικά βιώσιμη αλία. Ελπίζω πραγματικά η κοινή αλλιευτική πολιτική και η μεταρρύθμισή της να οδηγήσει σε μια αυθεντική αναγέννηση της όλης ε, αλλιευτικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τι θα έπρεπε να είχαμε μάθει. Υπάρχει ένα νέο βιβλίο το οποίο το αναφέρει ρητός. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται ε, ε ονομάζεται «Διαχείριση της αλληλείας, αποτυχία της πανδημίας και ε, εφικτές λύσεις». Το βιβλίο λέει ότι η διαχείριση των ελευμάτων κατά τη δεκαετία του 80 ήταν ε, αναποτελεσματική σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ήταν παγκόσμιο. Ποιες ήταν οι μέθοδοι αλληλείας είναι η λεγόμενη έλεγχη των εισρωών. Δείτε λίγο την εικόνα που έχετε εδώ στα δεξιά σας. Αυτό είναι ένα σύγχρονο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο είναι γεμάτο υπολογιστές, ε, ανιχνευτές αλευμάτων, ε, GPS και διάφορα άλλα μηχανήματα. Εκτιμάται ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ελίευση μας δίνει 5% περαιτέρω πιθανότητες να ε, αυξήσουμε τα λεύματά μας και αυτό αυξάνεται εδώ και δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία και με τα μικρά, ακόμα και με μικρά σκάφη, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιβιώσει αλληλεία. Θα αυξηθεί και θα φτάσουμε στην υπεραλίευση που έχουμε και τώρα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ σημαντικές συνέπειες ως προς τη διαχείριση. Γιατί λοιπόν δεν αρέσει το τρέχον σύστημα διαχείρισης των αλλιέων. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν τους αρέσει. Θα ήθελα να προσπαθήσω να μας ξυπνήσω από το λίχαρδο, λίχαργο με μία ρίση του Ντόν Πίβα που μάλιστα τα είπε αυτά τα πράγματα πριν από 45 χρόνια και μας έδωσε μια εικόνα του πώς θα ήταν ε, τα τρέχοντα συστήματα κανονισμοί αλληλεία για έναν άλλο τομέα, για την υλοτόμηση. Να σας δώσω εδώ τους κανόνες. Η υλοτόμηση θα επιτρέπεται τις Τρίτες και τις Παρασκευές ε, ε, και θα υπόκειται και σε περιορισμούς από διάφορες ανακοινώσεις. Θα είναι παράνομα για τον οποιονδήποτε εταιρεία, άτομο ή επιχείρηση να χρησιμοποιήσει ε, πριόνια ε, ηλεκτρικά για να ε, κόψει, για να λιτομήσει δέντρα. Τα κονοφόρα δέντρα θα μπορούν να κόβονται μόνο πριν από την 31η Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα εδώ. Οι αλληλείς είναι κυρίως επιχειρηματίες και η αλληλεία είναι μια νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα και όπως όλες ε, οι θέσεις εργασίας είναι ένας τρόπος ζωής, ε, μια νοοτροπία ζωής και είναι τμήμα και του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρωτίστως είναι επιχείρηση. Και αυτό σημαίνει ότι η αλληλεία ανταποκρίνεται στα ίδια κίνητρα στα οποία ανταποκρίνονται οι μικρές επιχειρήσεις. Και παρά την ε, ανεξαρτησία τους, οι αλληλείς ανταποκρίνονται στα κίνητρα και έχει αποτύχει η διαχείριση της αλληλείας ακριβώς γιατί σε μεγάλο βαθμό αγνοούμε αυτό το γεγονός. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι εμπορικές δυνάμεις να αντιμετωπιστούν και η πείρα μας μας δείχνει ότι αν περάσουμε σε ένα σύστημα ε, το οποίο θα ε, λαμβάνει υπόψη τα αλλιεύματα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Στους αλλιείς δεν αρέσει ε, να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα, θέλουν να έχουν αυτόν τον αγώνα για το ποιο θα πιάσει το, ε, το ψάρι, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον για αυτούς. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι όμως για να μειώσουμε το κόστος και σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς θα μείνουν εκτός δουλειά, διότι έχουμε υπεραλίευση στον τομέα της αλίας. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα νέο σύστημα. Οι αλληλείς δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ να συμμετάχουν στη διαδικασία διαχείρισης που μόλις σας περιέγραψα. Θεωρούν ότι είναι ένας ε, πατερναλιστικός ε, τρόπος ελέγχου και ε, χρησιμοποιούνται μέθοδοι εποπτείες και προσπαθούν να δούνε πώς μπορούν να κερδίσουν το σύστημα και να παρακάμψουν τους κανόνες. Τι θα κάνει λοιπόν τους αλληλείς να θέλουν να συμμετάσχουν πραγματικά σε ένα σύστημα. Η πείρα μας από όλο τον κόσμο υποδηλώνει ότι χρειαζόμαστε συστήματα τα οποία θα βασίζονται στα δικαιώματα. Και γιατί αυτό. Διότι όταν οι αλληλείς ε, έχουν συγκεκριμένο αριθμό μερίδιο του μέγιστο επιτροπόμενου αλλιεύματος, το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι περικοπές ε, γιατί θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους. Αν έχουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν χρησιμοποιούμε συστήματα δικαιωμάτων. Διότι υπάρχουν πάρα πολλέ λανθασμένες αντιλήψεις για τα συστήματα τα οποία βασίζονται στα δικαιώματα Αντίθετα με τα όσα λέει ο τύπο ε, για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, το να έχουμε τέτοια συστήματα δεν περιορίζονται σε συστήματα τα οποία ε, μεταφέρονται ατομικά ή έχουμε ITQ ε, συστήματα. Υπάρχουν διάφορα θέματα ε, περιφερειακά, ομαδική χρήση δικαιωμάτων και υπάρχουν υπέρ και κατά σε κάθε περίπτωση. Προκύπτει λοιπόν σαφώς αυτή τη στιγμή ότι η ιδέα το να έχουμε πλήρη δικαιώματα ε, ιδιοκτησία στην αλληλεία πραγματικά αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι θεωρητικώς αυτό θα μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ε, η ιδέα των ιδιωτικών συστημάτων ανταλλαγής δικαιωμάτων δεν θεωρείται κάτι το οποίο είναι σωστό. Ε, θεωρείται ότι είναι πολύ κακό όταν δίνονται τέτοια δικαιώματα και από την αλληλεία, αλλά η ιδέα να είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένα αυτά τα δικαιώματα δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ε, δεν θεωρούν ότι είναι μια πρακτική λύση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να περάσουμε σε αυτά τα συστήματα σε καμία περίπτωση. Το να υπάρχουν δικαιώματα, έστω και με ατέλειες, ε, είναι πολύ καλύτερο από το να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα ή να είναι πολύ αποδυναμωμένα. Ε, ωστόσο, ε, για λόγους αποτελεσματικότητας, για λόγους πρακτικούς, ε, η πλήρης ιδιωτικοποίηση των αλληλευτικών δικαιωμάτων δεν είναι πιθανό να συμβεί ακόμα και σε χώρες που είναι μακρά η παράδοση της αλληλείας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ισορροπία ώστε οι αλληλείς να μπορούν να διαχειρίζονται τους πόρους. Το συστήμα των δικαιωμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά το κράτος διατηρεί σαφή δικαιώματα για τους πόρους και δίνει μακροπρόθεσμη δυνατότητα χρήσης δικαιωμάτων, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση πλήρης ε, ιδιωτική ιδιοκτησία. Η πρόκληση είναι να έχουμε συστήματα τα οποία θα βασίζονται σε δικαιώματα, τα οποία θα αντικατοπτρίζουν τι συνθήκε, του κανόνε και τι δομέ διαχείριση που οι συμμετέχοντε και οι κοινωνικοί του θεωρούν ένομα και αποδεκτά. Επιπλέον θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουμε ως προς τη μετάβαση, την, την απασχόληση, τη δυνατότητα διαβίωσης και το τι ακριβώς θα γίνει όταν θα έχουμε συστήματα που θα βασίζονται στα δικαιώματα και θα εφαρμόζονται στην αλληλεία όπου υπάρχει ήδη υπεραλάβηση και υπερβολική χρήση των αποθεμάτων. Οι αλληλείς και οι κοινότητές τους λοιπόν θα μπορέσουν να έχουν οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν κυρίες και κύριοι. Τι μέλη γενέστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρτάται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Μπορούμε να συνεχίσουμε την άγουσα της υπεραλίευσης, υπερεκμετάλλευσης ε, και να ε, μειώνουμε την προσπάθεια ή μπορούμε να λάβουμε τη σκληρή πολιτική απόφαση να οδέσουμε προς μια αλληλεία στην οποία δεν θα έχουμε υπεραλίευση, δεν θα βασιζόμαστε σε ε, κανόνες ε, τύπου υλοτόμησης και θα επιτρέπουμε στους αλληλείς να έχουν την ελευθερία να λαμβάνουν αποφασίσεις που θα είναι αποδοτικές τους προς το κόστος επιχείρησής τους. Η επιλογή επαφείται σε εσά από εκεί και πέρα. Η ανάγκη να έχουμε μια καλή διαχείριση αλληλείας ε, γίνεται παγκόσμια πλέον. Δεν θα πρέπει να ε, βασιζόμαστε μόνο ε, στην διαχείριση από πάνω προς τα κάτω, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και οι αλληλείς. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την αλληλεία ώστε να συνεισφέρει στην ε, μείωση της ένδυας και στην ασφάλεια των τροφίμων και θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε ένα ουδέτερο φόρουμ για την υποστήριξη, ενθάρρυνση, επικοινωνία και την εκπαίδευση όλων μας για την υπεύθυνη αλληλεία. Θέλουμε να έχουμε ένα κόσμο στον οποίο η υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση της αλληλείας και οι πόροι της υδατοκαλλιέργειας θα είναι μεγάλη συνεισφορά στην ευημερία των ανθρώπων, στην ασφάλεια των τροφίμων και στη μείωση της ένδυας. Και τέλος, με τα κατάλληλα μέσα, η αλληλεία μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, σας ευχαριστούμε κύριε Βαλτιμάρσον. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίασή σας και σημειώνουμε με προσοχή όλα όσα μας είπατε. Είμαι βεβαία ότι θα σας υποβληθούν και πολλές ερωτήσεις μετά στη συζήτηση. Και πάλι για ένα τέταρτο δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Χέιρουπ. Χέιρουπ. Δεν καταφέρνω να το προφέρω σωστά, λέει ο Πρόεδρος. Καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο Ιχθιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης ε, στη Δανία. Έχετε το λόγο, κύριε Χέιρουπ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, θέλω να μιλήσω για διάφορες απόψεις της ε, αλληλείας. Από την ώρα όμως που το ψάρι ε, ψοφάει αρχίζει η αποσύνθεση του, του ο κρέατός του και ε, γι' αυτό ε, ε, προτιμούνται τα νοπά ψάρια, φρέσκα ψάρια. Υπάρχει λοιπόν διαφορά μεταξύ των, των ψαριών κατηγορίας Α και Β, δηλαδή αυτό που έχει αρχίσει από σύνθεση ε, των, ε, του σώματός τους. Ε, το ψάρι που εισάγεται στην Ευρώπη είναι η συνήθως ποιότητος Α ε, από χώρες όπου μπορεί να αγοραστεί φθηνά. Δηλαδή όσο πιο φθηνά αγοραστεί το ψάρι στην τρίτη χώρα τόσο πιο μεγάλο θα είναι το κέρδος κατά τη διακίνησή του στην Ευρώπη και ε, στην Ευρώπη διεξάγεται αλληλεία υψηλής ε, αξίας. Αυτά ξεκίνησαν από την βιομηχανοποίηση στην Ευρώπη, διότι προηγουμένως τα νοπά ψάρια υπήρχαν μόνο στην ε, ε, τοπική αγορά. Τώρα όμως είναι δυνατόν να υπάρχει ε, ψάρι πρώτης κατηγορίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και στο μέλλον θα μπορεί να υπάρχει παράκτη αλληλεία η οποία θα τροφοδοτεί όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά τώρα με αυτό πρέπει να μας απομακρύνει από την ιδέα ότι η αλληλεία πρέπει να βιομηχανοποιηθεί και αντιθέτως θα πρέπει οι περιορισμένοι αλληλευτικοί μας πόροι ε, να ε, ε, επικεντρωθούν στην πρώτη ποιότητα για να υπάρχει καλύτερη ποιότητα για τον καταναλωτή και μία αηφόρος οικονομία για τις αλλιευτικές κοινότητες της Ευρώπης. Υπάρχουν διάφορες μορφές της αλληλείας, καταρχήν ε, με ε, πλοία στην ανοιχτή θάλασσα όπου επικεντρώνονται σε αλληλευτικές περιοχές όπου μπορούν να επικεντρώσουν όλα τα μέσα τους και μπορούν να βρουν μεγάλη συγκέντρωση ψαριών. Και εδώ το μέγεθος του ψαριού είναι πολύ σημαντικό και πρέπει επιπλέον να μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί το ψάρι σε μεγάλες ε, αποστάσεις. Στο παρελθόν υπήρχε ε, μόνο υπήρχαν μόνο αλατισμένα ψάρια από μακρινές περιοχές ενώ ε, τα νοπά ψάρια ε, προέρχονται από την παράκτιο αλληλεία γύρω στην Ευρώπη και ε, υπήρχε μία διέρεση μεταξύ των περιοχών κατά τρόπον ώστε ο κάθε ένας, ο, η κάθε οικογένεια, ο κάθε ψαράς να έχει την συμμετοχή του. Ε, για να μπορέσει να διατηρηθεί και το ενδιαφέρον. Αυτό το ψάρι ε, πωλείται την ημέρα που αποβιβάζεται και τροφοδοτεί ε, την ποιότητα αλφα ψαριού στην Ευρώπη. Γύρω στο 1900 ήταν κατέστη δυνατόν η, τα παράκτια, η παράκτια να επενδύσουν σε όλο και μεγαλύτερο καλύτερα σκάφη και ε, να ε, επικεντρωθούν σε ταξίδια πολλών ημερών μακριά από τις ακτές για βιομηχανική ε, αλληλεία και μεταξύ του 1900 και του 2000 αυξήθηκε αυτή η αλληλεία ανοιχτής θαλάσσης. Δεν μπορούσε όμως να φτάσει στην Ευρώπη γέρο και να επιτύχει την επιζητούμενη αξία και γι' αυτό χρειάστηκε ε, να αναπτυχθεί ολόκληρη υποδομή. Τα διάφορα δίκτυα τα οποία έχουν δημιουργηθεί έχουν ενταχθεί και στην εσωτερική αγορά και στο ε, μέλλον ακόμη τα ψάρια πρώτης κατηγορίας θα έχουν μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Δηλαδή οι δανέ Κινέζοι μπορούν να τροφοδοτήσουν 7 ευρωπαϊκά εστιατόρια και ε, να υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα η οποία να έχει την δυνατότητα να επικεντρωθεί εις, ε, την αλληλεία η οποία οφείλεται εις ε, το αλίευμα να μπορεί να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση ε, και χρησιμοποιούνται διάφορα ελγαρία, πρόκειται για πλοία με μικρές μηχανές και λίγη κατανάλωση πετρελαίου ε, χωρίς να καταστρέφουν το υπέδαφος ε, και την παραγωγή και τα αλλιευτικά μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες. Τα μεγάλα αλλιευτικά που ψαρεύουν ψάρια πρώτης κατηγορίας ε, και ε, τα μικρότερα τα οποία έχουν έχουν επικεντρωθεί ε, στην κατηγορία ε, ε διότι ε, και οι μεγάλοι εξοπλισμοί μπορούν να βλάψουν την ποιότητα του ψαριού. Το σύστημα σήμερα είναι ολοκληρωμένο αλλά προβληματικό. Ε, υπάρχει χρήση βιομηχανικών ε, μέσων για να επιλύσουμε ε, ορισμένα προβλήματα αλλά οι εξελίξεις στην Ισλανδία είναι πολύ χαρακτηριστικές. Είδαμε ότι το 2003 και το 2007 ανεπτύχθη ένα τομέα ή στην ε, Δανία όπου οι ιδιωτικές τράπεζες και οι τράπεζες που χρηματοδοτούν την αλληλεία είχαν διαθέσει υπερβολικές πιστώσεις ε, και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ζημίες τους έδιναν ε, λοιπόν εις τα πλοία όχι όμως εις τα πλοία πληρώματα, ιδιοκτησία των ποσοστώσεων αλίες για να προσπαθήσουν να μειώσουν τον αριθμό των πλοίων, δηλαδή οι τράπεζες τερικά είχαν στα χέρια τους τις ποσοστώσεις και κατόπιν αυτού τα μικρά πλοία κατανάλογαν μεγαλύτερες ποσότητες ποσοστώσεων και τα μεγαλύτερα πλοία δεν είχαν τη δυνατότητα να ψαρεύσουν στο επίπεδο των αναγκών τους. Υπήρχε η δυνατότητα λοιπόν να πολιθούν αυτές οι ποσοστώσεις και ε, πολλές, ε, ε, πολλά πλοία μπόρεσαν ε, να μεταφέρουν τις ποσοστώσεις άλλων στα δικά τους, ε, ε, δικά τους πλοία και μονοπόλησαν τις ποσοστώσεις χρησιμοποιώντας τους σαν δικιά τους ιδιοκτησία. Αυξήθηκαν λοιπόν οι τιμές για τις ποσοστώσεις πελαγίσιων ψαριών πάρα πολύ διότι ε, υπήρχε μία εγγραφή των εταιριών σαν ε, ε, στα αλλιευτικά στους αλλιευτικούς καταλόγους για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ποσοστώσεις οι οποίες του διδυνόντουσαν για να κερδίσουν ε, δια της πωλήσεώς τους ε, και χρειάστηκε μία αστυνόμευση των ποσοστώσεων καθότι το πρώτο χρόνο 25% των πλοίων στη Δανία που αλλιευάν ε, εξαφανίστηκε και είδαμε ανταυτού μεγάλα πλοία μόνο που είχαν ευξημένες δυνατότητες και τα οποία εξαρτώντουσαν από τις τράπεζες. Κατόπιν αυτού ε, εξαφανίστηκε ένα μεγάλο μέρος της αλίες, ε, πράγμα το οποίο ε, δυσχέρανε την κατάσταση για τα πληρώματα και είχε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Ορισμένοι έγιναν πολυεκατομμυριούχοι, ενώ άλλοι έχαναν τη δουλειά τους, ακόμη και αν στο παρελθόν είχαν ψαρέψει μαζί όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο, κάποιος ασχολείται ακόμη με αυτόν τον τομέα είναι κάποιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις ποσοστώσεις και προσπάθησε ε, είτε ε, να ε, εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες ποσοστώσεις του είτε να τις πουλήσει σε νεότερους αλληλείς οι οποίοι δεν είχαν ποσοστώσεις. Ε, οι περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα αποθέματα αλλιές είναι οι πιο επιζητούμενες και ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει κανείς την τιμή του ψαριού το οποίο αποβιβάζεται και ε, οδηγεί σε ποσοστώσεις αλλιεύσεως και όχι αποβίβασης ενώ στο παρελθόν υπήρχε ένα προηγούμενο σύστημα. Το σύστημα αυτό ενθαρρύνει αυτή την ανήθικη συμπεριφορά ορισμένων ψαράδων και έχουν δημιουργηθεί συγκροτήματα όπου ε, ε, ενοικιάζονται οι αλληλείς που δεν έχουν ποσοστώσεις για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση του ελευτικού στόλου. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ε, υποβάθμιση ε, του των ποσοστώσεων εάν υπήρχαν, ε, υπήρχε μια συγκέντρωση των ποσοστώσεων όπου οι ποσοστώσεις ναι μεν ε, θα ανήκαν στο κράτος αλλά θα αποδίδονται σε εγγεγραμμένους ε, αλληλείς οι οποίοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλλιέων αντί ε, να υπάρχουν μονοπόλια. Στην ε, Δανία υπάρχει μια σοβαρή οικονομική κρίση αυτή την εποχή και χρειάστηκε να αναπτυχθεί η παράκτη αλληλεία ε, για να υπάρξουν επαρκείς ποσοστώσεις. Τώρα όμως οι ποσοστώσεις αποφασίζονται ιδίως από τους τραπεζίτες. Ε, και βλέπετε εδώ ότι ε, η ομάδα των αλλιέων έχουν μειωθεί πολύ διότι οι παράκτη αλληλείς μπόρεσαν και κατήρτισαν μία στρατηγική η οποία τους επιτρέπει να αποβιβάζουν τα, πλοία, τα ψάρια τους ως αλλιεύματα πρώτης κατηγορίας και να διατηρήσουν τα δικαιώματα αλίας σε ένα κοινό συγκρότημα αντί ο ένας να πουλάει τα, ε, τις του ή στον άλλον ε, αυτά συνέβησαν μέχρι την άνοιξη του 2007 και στη συνέχεια οι αλληλείς διαχειρίστηκαν μόνοι τους τις, τα αλλιευτικά δικαιώματα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία σταθερή τιμή η οποία πληρώνεται από κάθε μέλος του συνεταιρισμού για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις και ε, στο τέλος ε, καθορίζεται και το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις τράπεζες για την αποπληρωμή των δανείων βλέπουμε ότι ε, είναι μια κοινότητα η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τους πόρους της ε, και ε, στο μέλλον αποβλέπουμε σε, στην βιολογική αλία βλέπουμε όμως ότι εάν οι τιμές των ε, ποσοστώσεων είναι αστρονομικές τότε ε, ε, υπάρχει χρεοκοπία και γι' αυτό οι εταιρείε χρειάστηκε να παλέψουν για να επιβιώσουν μέσα στις κοινότητές τους και πριν εισαχθεί το νέο σύστημα δεν χρειαζόταν η μέθοδοι αυτή μπορούσαν να να διαχειριστούν τις ε, διακυμάνσεις στην αλληλεία και υπήρχε μια ισχυρή κοινότητα ενώ τώρα ε, 100 ε, ε, εκατομμύρια κορώνες είναι το διακύβευμα το οποίο ρυθμίζεται από τις τράπεζες οι οποίες αποβλέπουν οι σκερδοσκοπικές αγορές ενώ υπάρχει μεγάλη κρίση στον αλληλευτικό χώρο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ε, την δημιουργία των ε, των ε, συγκροτημάτων για να μπορέσει ε, να υπάρξει ε, καλύτερη αριεία και οι εταιρείε, ε, τα συγκροτήματα αυτά εταιριών θα ε, πρέπει να έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για να ανανεώσουν, να ανανεώσουν το στόλο τους και υπάρχει υπάρχει ε, ένα ε, ποσοστό ε, αλληλείας ποιότητος α το οποίο πρέπει να καλύπτει το 80% του συνόλου και να αναφέρεται εις έύματα τα οποία δεν απέχουν πέραν των 24 ώρων από την κατανάλωση. Κατά αυτόν τον τρόπο οι τοπικές ε, ομάδες θα μπορούσαν ε, ε, να αγοράσουν ποσοστώσεις και αλλιευτικά δικαιώματα και ε, θα χρειαστεί ε, στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπον ώστε οι ποσότητες οι οποίες ε, διανύμονται να παραμείνουν στα όρια της αηφορίας των ειδών. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα προβλήματα της βιομηχανικής αλληλείας διότι εάν προωθήσουμε την παράκτη αλληλεία θα έχουμε καλύτερης ποιότητας ψάρια. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν θα ήθελα να ξεπεράσετε το τέταρτο που έχετε στη διάθεσή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φρέντρικ Λουντμπερκ που είναι πρόεδρος της Οργάνωσης Ελιαίων των νησιών Όλαντ, που βρίσκονται μεταξύ Φιλανδίας και Δανία. Έχετε το λόγο. Ονομάζομαι Φρέδρικ Λούντμπερκ και εκπροσωπώ εδώ τα νησιά Όλαντ, δηλαδή την οργάνωση αλλιών των νησιών Όλαντ. Τα νησιά Όλαντ είναι μια πολύ μικρή περιοχή στη Βόρεια Βαλτική. Απαρτίζεται από 27.000 κατοίκους και 250 εγγεγραμμένους αλλοίς με πάνω από 300 σκάφη, 90% των οποίων χρησιμοποιούνται για παράκτη αλία. Θα σας μιλήσω εδώ για την συντήρηση των πόρων και την διαχείριση του ελευτικού στόλου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ε, μικρής παράκτειας αλίας. Έχουμε μία μοναδική θέση στη Βαλτική θάλασσα, γιατί είμαστε αυτοδιαχειριζόμενοι σε πολλού τομεί, ε, μεταξύ άλλων και στην Αλία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε το δικό μα νόμο στην Αλία, που μπορεί να ε, διαφέρει τελείω από την αληφτική πολιτική τη Φιλανδία, στην οποία ανήκουν ε, τα νησιά Όλαντ. Η, Αλία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κλάδο των νησιών Όλαντ. Και νομίζω ότι γνωρίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, για την ευδοκίμηση της μικρής παράκτειας αλίας. Η μικρή παράκτεια αλία είναι πολύ σημαντική για τη ζωή των νησιών Όλαντ. Μάλιστα, είμαστε και από το 1995 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πλούσια εμπειρία από την εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και είδαμε τις συνέπειές της στην αλληλεία μας. Και αυτή την εμπειρία θα ήθελα να σας μεταφέρω εδώ και να τη συζητήσουμε. Θεωρούμε ότι η παράκτη αλληλεία ανταποκρίνεται σε ένα, μια ειδική δέσμη προκλήσεων που μέχρι στιγμής δεν ελήφθησαν υπόψη στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Για παράδειγμα, η παράκτη στο όλοι έχουν ε, τεράστια ε, ε, εμπορεύματα σε σχέση με άλλου είδους αλία. Δηλαδή, εμείς τα ψάρια που πιάνουμε θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και αλλιώς, πέραν της αλίας. Και μάλιστα προσπαθούμε λιγότερο ψάρι να έχουμε μεγαλύτερη κερδοφορία διαθέτοντας τα ψάρια αυτά στην αγορά. Μερικές φορές έχουμε άμεση διάθεση προς το καταναλωτή. Και μάλιστα η προσαρμοστικότητα του των αλλιέων στην, στις ανάγκες της τοπικής αγοράς είναι πολύ σημαντική. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι ελευτικές δυνατότητες υπάρχουν και τι επιλογές. Πάντως αυτό που είναι σωστό για τη μικρή παράκτη αλία η για όλα, Όλαντ ίσως έχει ελεύθερο αποτέλεσμα σε άλλες περιοχές. Πάντως θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στους τοπικούς παράγοντες, στους τοπικούς επιχειρηματίες ε, να κάνουν τις επιλογές τους. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια νέα πολιτική με ένα κοινό νομικό πλαίσιο εξαιτία των ιδιαιτεροτήτων, αλλά και επειδή είναι πολύ χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλού περιορισμούς και απαγορεύσεις που περιορίζουν την παράκτεια αλία. Κάτι που παραβλάπτει και τι επιδόσει ε, του στόλου τη παράκτεια αλίας. Θα αναφερθώ αργότερα στι συνέπειε που έχει η κοινή πολιτική στη αλία μα, αλλά θα ήθελα να υποβάλω κάποιε προτάσει. Είναι απλούστατε οι προτάσει αυτέ. Γνωρίζουμε ότι ο πιο κατάλληλο για να λάβει τι αποφάσει ε, για την αλία στα δικά μα ύδατα είμαστε εμεί ίδιοι. Και το γνωρίζουμε αυτό γιατί αυτή ήταν η πολιτική μα ε, για αιώνε. Τα τελευταία 15 χρόνια όμω, από τότε που ενταχθήκαμε στην κοινή αλληλευτική πολιτική, είδαμε τις επιδοτήσεις ε, που οδήγησαν σε μείωση των αλληλευτικών, των ε, αποθεμάτων και επηρέασε την κατάσταση παράκτη αλίας. Επίσης, η δυσπιστία των αλίαων και του κοινού προς τα αλλιευτικά προϊόντα είναι χαρακτηριστική. Γνωρίζω ότι Ίσως οι προτάσεις μου φαίνονται κάπως ε, ριζοσπαστικές, αλλά δεδομένου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αλία μας, νομίζω ότι είναι ευνόητο ότι υποβάλλουμε τόσο ριζοσπαστικές προτάσεις. It is very important that you understand... Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι η παράκτη αλία είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η παράκτη αλία στη, στο Σουδικό Αρχιπέλαγο, στη Βαλτική, που είναι παρόμοιο με το δικό μας το νησιόν Όλαντ, δεν είναι αλία μικρής κλίμακας. Εμείς αλληλεύουμε κυρίως ελευθερικά είδη που δεν εμπίπτουν στις ε, αλλιευτικές ποσοστώσεις. Επίσης η αλληλεία μας είναι κυρίως εποχιακή για τα θαλάσσια είδη, όπως είναι ο Σολομός ε, και μερικές φορές ο Γάδος. Ο Γάδος είναι πολύ σημαντικός για μας γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν θετικές συνθήκες, κάτι 25 με 30 χρόνια, για μια άνθηση του ελευτικού είδους του γάδου. Στην δεκαετία του 70 και 80 είχαμε τέτοια άνθηση του γάδου. Τότε επικρατεί στην παράκτη η ελία γάδου. Ενώ άλλες φορές ε, τον υπόλοιπο καιρό ελιεύουμε αλευτικά είδη που δεν εμπίπτουν στα τάκ. Επίσης έχουμε παράγωγη ελία, προσπαθώντας να αλλιεύσουμε γάδο. Βέβαια αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινή αλλιευτική πολιτική που περιόρισε δραστικά την αλία Για να χρησιμοποιήσουμε όμως το γάδο όταν αρχίζει η αλλιευτική περίοδος πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα αλλιευτικά αποθέματα, στους αλλιευτικούς πόρους. Και με την σημερινή κοινή αλλιευτική πολιτική δεν έχουμε τέτοια πρόσβαση. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική στην παρακτέλεια. Δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία ή έρευνα στα θέματα αυτά, αλλά τι τελευταίε δεκαετίε που ασχολούμαι με την παράκτη αλεία προσπάθησα να εντοπίσω τα συστατικά της επιτυχίας τη παράκτη αλίας. Μερικοί έχουν καταφέρει να βρουν αυτά τα συστατικά και άλλοι όχι. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει κανεί ποια είναι η ακρογωνία λύθη τη επιχείρηση και ποιε είναι οι συνθήκε οι κατάλληλε συνθήκε για την παράκτη αλία. Οι ελευτικές δυνατότητες είναι το ένα στοιχείο. Βέβαια εξαρτάται από το αλληλευτικό είδος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε όμως σε αυτές τις αλληλευτικές δυνατότητες, γιατί μπορεί από φυσικούς λόγους ή από διάφορες οικολογικές διακοιμάσεις να μην έχουμε σταθερές αλληλευτικές δυνατότητες. Επίσης υπάρχουν κάποια φυσικά εμπόδια στην κατάσταση της, της παράκτης αλίας. Πάντω, ε, ένα από τα θεμέλια τη παράκτη ελίας που μπορούμε να το διαχειριστούμε είναι τα εμπόδια από την ε, πολιτική και την ομοθεσία. Αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε και γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα για να σα αναπτύξω αυτό το θέμα. Και το τελευταίο θεμέλιο τη κατάσταση ε, τη παράκτη ελίας και το πιο σημαντικό είναι οι επιχειρηματικέ ευκαιρίε για τον κλάδο της παράκτη ελίας. Οι ελίες που κατάλαβαν τη σημασία της επιχειρηματικής προοπτικής είναι πολύ επιτυχημένοι επαγγελματίε. Παρόλο που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, παρόλο που δεν συντρέχουν πάντα όλα τα θεμέλια, αυτοί οι τέσσερις λόγοι που σας ανέφερα. Και εδώ είναι οι ελευτικές ευκαιρίες ε, της περιοχής ε, των νησιών Όλαντ. Έχουμε αρκετά καλές ε, ελευτικές δυνατότητες για ελευτικά είδη που δεν εμπίπτουν στα ΤΑΚ και τα πιο σημαντικά επειδή, ακριβώς επειδή είναι επίπτωση στα τάκ, δεν επηρεάζονται αυτά τα ίδια από την αλληλευτική πολιτική. Ο στόλος μας είναι πολύ ευέλικτος, επειδή ακριβώς αλληλεύει παράκτη και πολλές φορές ε, εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Τα, βέβαια πολλά αλληλευτικά ύδατα είναι ιδιωτικά και αυτό είναι δύσκολο ως προς την πρόσβαση. Γιατί ο ιδιοκτήτης τους έχει το δικαίωμα να αλληλεύει εκεί. Αυτό είναι ένα φυσικό εμπόδιο φυσικά στην Αλία, το, η ιδιωτική ιδιοκτησία των υδάτων σε πολλά σημεία. Αυτό είναι ένας χάρτης των νησιών Όλαντ, μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας και βλέπετε την κόκκινη γραμμή και ποια τμήματα είναι ιδιωτικά. 90% της ε, αλίας γίνεται εντός ε, της κόκκινης αυτής γραμμής. Μακάρι να μπορούσα να σα δώσω περισσότερε πληροφορίε για τον τρόπο διαχείριση τη αλληλεία στα νησιά Όλαντ. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, επιτύχαμε τουλάχιστον στα αλληλευτικά είδη που δεν ανήκουν, δεν εμπίπτουν στα ΤΑΚ, μια αηφόρο διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Όταν βρίσκεται κανεί στη Βόρεια Βαλτική, αντιμετωπίζει πολλά φυσικά εμπόδια. Καιρό, άνεμο, πάγο για παράδειγμα. Η παράκτη αλληλεία είναι στο έλεος του καιρού Πολλά δε μάλλον που ασκείται με μικρά αλληλευτικά σκάφη. Έχουμε τεράστιες ζημίες από τις φώκες και από τους κορμοράνους. Επίσης έχουμε άνθηση των, των φυκιό, φυκών εξαιτία της ευτροφίας στη Βαλτική θάλασσα, που καθιστά δύνατη μερικές φορές την αλληλεία. Και η γενική κατάσταση Βαλτικής δεν ε, ευνοεί την αλία ούτε των ειδών που εμπίπτουν σε τάκη, ούτε των ειδών που είναι εκτός των αλληλευτικών ποσοστώσεων. Μία χαρακτηριστική εικόνα, πάνω από 50% των ψαριών που αλλιεύονται με απλάδια ε, γίνονται βορρά των, των φωκιών. Είναι μια κατάσταση που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι αλληλείς στα υδατά μας. Επιχειρηματικές ευκαιρίες που είναι ακρογωνιαίος λήθος ε, της αλληλείας και δυστυχώς ε, όχι αρκετά ανεπτυγμένο. Οι Ελλείς πια δεν περιορίζονται στην αλεία, αλλά θέλουν να έχουν μια κερδοφόρο απασχόληση από τα ψάρια που αλλιεύουν και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εδώ διεξόδου επαγγελματική και επιχειρηματική για τους Ελλείς. Και αυτό ήταν ένα πολύ δύσπεπτο μήνυμα για τους Ελλείς. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν ονοτροπία και να αλλάξουν πλήρω την προσέγγιση του ελευτικού επαγγέλματο. Οι αλλοί πια αρχίζουν και γίνονται περισσότερο επιχειρηματίε παρά αλλοί. Κάτι που είναι απαραίτητο για να επιτύχουν στην δραστηριότητά του. Πρέπει να γίνει μια μεταβίβαση και μετάβαση και προ την επιχειρηματικότητα. Όπω σα είπα, είναι μικρό, μικρή ποσότητα των ψαριών που αλλιεύουμε, γι' αυτό και χρειάζεται μια ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματο, ιδιοχέτευση στην τοπική αγορά, Οπότε υπάρχει προστιθέμενη αξία με τη μεταποίηση του αλλιεύματος, τη φιλετοποίηση, το καθαρισμό κτλ. Και πρέπει να συνδυάζεται η εποχιακή αλλία με μερική ή πλήρη απασχόληση. Αυτές είναι μερικές από τις επιχειρηματικές διεξόδους που έχουν οι Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να σας περάσω με την ομιλία μου. Υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια και κολλήματα από την πολιτική και την νομοθεσία και υπάρχουν και τόσα άλλα προβλήματα για τους ελλείς που καλό θα ήταν να αποφευθούν τουλάχιστον αυτά τα εμπόδια που δημιουργούν η νομοθεσία και η πολιτική. Θα πρέπει να μπορούμε να λιεύουμε όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. Βέβαια, είναι κάπως αναλαστική η νομοθεσία, δεν μπορούμε να αλλάζουμε αλλιευτικά εργαλεία, υπάρχει ο περιορισμός των ποσοστώσεων, υπάρχουν οι κλειστές αλλιευτικές περίοδοι, η συνεχής τροποποίηση της νομοθεσίας, μία στάθεια ό,τι αφορά την πρόσβαση στα ΤΑΚ. Όλα αυτά είναι νομοθετικά προβλήματα και προβλήματα πολιτικής. Και επιπλέον αυξημένοι αλληλευτικοί έλεγχοι οδηγούν σε μία αλλοπρόσελη και παράλογη γραφειοκρατία. Η παράκτη Ελία αντιμετωπίζει συγκεκριμένε προκλήσει. Δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί, έχουμε μαζικές μερικές φορές μερικές μαζικές αλλιεύσεις και πρέπει να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και να αυξήσουμε την κερδοφορία με μικρό, με λιγότερο ψάρι, γιατί είναι τεράστια και τα έξοδα της μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα μετάβασης σε διαφορετικό ελευτικό είδος και σε διαφορετικό ελευτικό εργαλείο, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η σημερινή ελευτική πολιτική έχει πολλές απαγορεύσεις και περιορισμούς και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις της παράκτιας αλίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούνμπερκ. Στη συνέχεια Έχουμε τη συζήτηση με τους ε, συναδέλφους. Ο κύριος Βαλέσσα ζήτησε το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι με την ακρόαση αυτή φτάνουμε στην καρδιά των προβλημάτων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μιλούμε για τη συντήρηση των αλληλευτικών πόρων, την ε, διαφύλαξη του οικοσυστήματος, τη διαχείριση του αλληλευτικού στόλου στο, στην πρώτη μιλία ακούσαμε για το οικοσύστημα και την συνεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των διαφθόρων αλληλευτικών ειδών. Επίσης μιλήσαμε για τη διαχείριση των στόλων. Η αλληλεία είναι πάνω απ' όλα οικονομική δραστηριότητα. Οπότε η λειτουργία της θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία οικονομίας της αγοράς που μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στο πρώτο σκέλος, δηλαδή στην διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Είπαμε ότι υπάρχει συνεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων αλλιευτικών πόρων και αποθεμάτων. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει μεταξύ της Αρδελόρεγκας και του Γάδου στη Βαλτική θάλασσα. Ο, ο, ο πρώτος, η πρώτη απειλή για τον ε, Μπακαλάο είναι η Σαρδελόρεγκα και όχι η Αλής. Όσο μεγαλύτερα είναι τα αποθέματα της Σαρδελόρεγκας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση προς τα αποθέματα του Γάδου. Βέβαια, πολλές φορές η κατάσταση αντιστρέφεται και μερικές φορές υπερέχουν τα αποθέματα του γάδου έναντι σαρδελόρεγας. Στα, στη δεκαετία του 70 είχαμε τα υψηλότερα αποθέματα γάδου και το αντίθετο στην Σαρδελόρεγκα. Και για πάλι έχουμε μια αναζωογόνηση των ε, αποθεμάτων γάδου στη Βαλτική εις βάρος των αποθεμάτων της ε, Σαρδελόρεγκας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση τώρα των αλληλευτικών πόρων έχουμε και άλλους παράγοντες που παίζουν ρόλο. Πολύ σημαντικό, πολύ είναι να υιοθετήσουμε μια οικοσυστημική προσέγγιση. Να έχουμε τον κώδικα της υπευθύνης αλίας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ε, νέα κοινή πολιτική. Και μάλιστα η γνώμη μας για τη συνεξάρτηση των διαφόρων θαλάσσιων οικοσυστημάτων ε, δεν είναι ακόμη πλήρης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε επιστημονικές μελέτες και επιστημονικά πορίσματα που θα στοιχειοθετούν ε, τις δικές μας προτάσεις. τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης είναι ένα πολύ σωστό βήμα και νομίζω ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να στραφούμε και να τη συνεχίσουμε. Βέβαια, όλα αυτά τα μακροπρόθεσμα σχέδια δεν είναι αμετάκλητα. Θα πρέπει, ούτε θα πρέπει να είναι αδιάλεκτα. Θα πρέπει να περιέχουν και κάποιο περιθώριο λιγμών, κάποια ελαστικότητα για να προσαρμόζονται καλύτερα στις αλλαγές και στο περιβάλλον, αλλά και στην κατάσταση των αλλιευτικών πόρων. Ο υπερβολικός περιορισμός των αλλιευμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των απορρίψεων ή σε απόκρυψη των αλλιευμάτων. Πάντως, ας μην ξεχνούμε ότι και η αλλιείς είναι τμήμα του οικοσυστήματος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς οι νέες νομοθετικές διατάξεις θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά των αλλιέων. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διαχείριση του ελευτικού στόλου. Το τεράστιο ελευτικό δυναμικό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ε, κοινοτικής αλίας. Αλλά ας μην ξεχνούμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η αλία είναι μια οικονομική δραστηριότητα και ένας μικρότερος ε, στόλος που δεν ε, θα υπάγεται στις αρχές της οικονομίας είναι το ζητούμενο για μας. Δηλαδή θέλουμε μια οικονομική δραστηριότητα να ακολουθεί οικονομικούς κανόνες, το ίδιο και η αλία. Μιλήσαμε σήμερα για την εισαγωγή του συστήματος ΙΤΕΚΟΥΜ. Έτσι διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του ελευτικού στόλου, μία βελτίωση της κερδοφορίας και οι κρατικές επιδοτήσεις για τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση του ελευτικού στόλου, με ταυτόχρονη απόσυρση παροπλισμό ενός τμήματός του. Επιπλέον, η εισαγωγή ορισμένων μέτρων στη Βαλτική θάλασσα δεν ε, είναι κατά ανάγκη κατάλληλη και σε άλλες αλλιευτικές λεκάνες. Η Πολωνία μείωσε κατά 40% το αλληλευτικό της δυναμικό και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται περιορίζεται όλο και περισσότερο. Το πρόβλημα όμως ε, έγκυται στην, στον εξυγχρονισμό του στόλου ελίευσης πελαγικών ειδών. Εκεί δεν ε, αξιοποιούνται όλες μας οι δυνατότητες. Καλό θα ήταν να διαβρυνθούν τα αλληλευτικά πεδία για να βελτιωθεί η αλληλευτική δραστηριότητα στην θάλασσα, κάτι που δεν επιτρέπεται από τις ε, νομοθετικές διατάξεις. Και εδώ λαμβάνει η χώρα μια διακριτική μεταχείριση για ένα τμήμα του πολωνικού αλληλευτικού στόλου. Γιατί οι παλιέ χώρε μέλη προσάρμοσαν το στόλο του στην αλία των πελαγικών ειδών σε προηγούμενε περιόδου, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Πολωνία. Και επαναρχόμενο στο σύστημα διαχείριση του ελευτικού στόλου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αλληλευτική εκστρατεία, εδώ δεν υπάρχει ιδεώδη λύση και ενιαία για όλου. Και το σύστημα αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά εμπεριέχει κάποιε απειλέ που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτού του συστήματος το θέμα το σύστημα αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνεται όχι μόνο από τις κοινοτικέ διατάξεις, αλλά και από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Και οι βασικές ε, αποφάσεις για τα θέματα αυτά θα πρέπει να επαφίονται στην ε, διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και τέλος, πραγματικά τέλος, θα ήθελα να πω ότι η μείωση του στόλου σχετίζεται και με τη μείωση της απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να θεσπίσουμε και κάποιους μηχανισμούς αντιστάθμισης σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια μείωση στόλου. Γιατί ούτω ή άλλω σε περιοχέ που στηρίζονται στην Αλία και πολλοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά του δεν υπάρχουν άλλε επαγγελματικέ διέξοδοι και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Βαλώσα. Ο κύριο Γκρόμπολτσικ. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω μία ερώτηση προς τον καθηγητή Τόμας Χόιρουπ. Μιλήσατε για την αλληλεία ειδών πρώτης κατηγορίας ή δεύτερης κατηγορίας Α, Α και Ε. Και είπατε ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος αλλήλευσης τέτοιων ειδών Α και Ε και οι συνέπειες διαφορετικές. Αλλά εσείς ε, μιλήσατε κυρίως για την ε, Βαλτική θάλασσα. Το 20% των αλλιευμάτων ε, αλλιεύονται με τέτοιο τρόπο, γιατί το 80% των αλλιευμάτων της Βαλτικής είναι βιομηχανική αλλιεία. Αλλιεία για δόλωμα, που δεν έχει καμία διαφορά αν είναι πρώτης ποιότητας ή δεύτερης ποιότητας, γιατί ουσιαστικά γίνεται μαζική αλία από τεράστια σκάφη με στόχο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αλλιεύματα ως ηχθιάλευρα. Οπότε η επιρροή αυτής της, αυτού του είδους ελιές, α, για Παρασκευή ηχθιαλεύρων, πώς επηρεάζει την κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων, γιατί αυτή είναι η μαζική αλία που γίνεται στη Βαλτική. Ο κύριος Λούντεμπερκ μίλησε για την παράκτη αλιά μικρής κλίμακας. Τι επιρροή είχε η θέσπιση των ποσοστώσεων ITQ στην περίπτωση της παράκτης αλίας. Ευχαριστώ. Eh, Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Η κυρία Λέβη. frågeställningen som herr kom med angående fiskmjöl och fisk, foderfiske i Ήθελα να κάνω και μία επιπρόσθετη ε, ερώτηση σχετικά με τα ηχθιάλευρα και ε, τις δραστηριότητες ε, τις αλλιευτικές στη Βόρειο Θάλασσα διότι είπατε ότι σύμφωνα με τη ΦΑΟ 45% των ψαριών τα οποία καταναλώνουμε είναι ε, ε, ε, ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το ποσοστό των πόρων που διατίθεται για, για να τραφούν αυτά τα τα ε, ψάρια της ε, ε, καλλιέργειας και επίσης θα ήθελα να ξέρω επειδή υπάρχουν ε, διαφορετικές πληροφορίες όσον αφορά τις ποσοστώσεις, ε, τι γίνεται. Ήταν πολύ θετικό να ακούσουμε ε, τι εικόνα θα είχαν αυτά τα ITQs, δηλαδή ότι δεν είναι η κατάσταση σαν την Ισλανδία όπου υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τα ITQ, διότι μεγάλοι επενδυτές αγοράζουν τις ποσοστώσεις και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να σκεφτούμε ότι το ψάρι στη θάλασσα ουσιαστικά είναι άγρια φύση και η ε, ε, φύση αυτή μας ανήκει σε μας και στις επόμενες γενιές. Οπότε πολύ σωστά λέγεται ότι το κράτος πρέπει να διατηρήσει δικαιώματα πάνω σε αυτούς τους πόρους και ιδίως η, ε, να μπορέσουν ε, να ε, ε, υπάρχουν ανανεώσεις ε, των ε, leasing τα οποία θα, τα είναι συνδεδεμένα με ορισμένα προνόμια για τη χρήση τους. Δηλαδή εάν θέλει κανείς να έχει πρόσβαση στην άγρια φύση θα πρέπει να, καλύπτει, να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μεθόδους ε, πιο θετικές και με τι κοινωνικά κριτήρια. Πέραν αυτού, θα έπρεπε να αποφύγουμε ε, κάθε κερδοσκοπία και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Βαλτεμάζερ. Έχετε σκεφτεί ότι ε, καταρχήν πρέπει κανείς να αγοράσει αυτά, ε, αυτές τις ε, αλλιευτικές άδειες. Δεν υπάρχει ελεύθερη χορήγηση και αυτό διατίθεται για μία δεκαετία αλλά πρέπει να συνεπιφέρει και ορισμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή αν κανείς υπεραλλιεύει, αν έχει βλαβερές επιπτώσεις ή στο οικολογικό σύστημα και στη θάλασσα δεν θα έπρεπε να πληρωθεί και κάποια αποζημίωση για τις ζημιές οι οποίες δημιουργήθηκαν και αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις της ξηράς. Αν δηλαδή οι ε, επιχειρήσεις στην ξηρά καταστρέψουν τη φύση είναι υπεύθυνε. Ε, για να υπάρχει λοιπόν σωστή διαχείριση της αλληλείας θα πρέπει επίσης να υπάρχει ε, μία υποχρέωση οικονομικής καλύψεως εάν υπάρξει κάποια ζημιά. Ευχαριστώ. Να θέσω και εγώ μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της ΦΑΟ. Είναι η εξή. Νομίζω ότι πολύ καλά μας εξηγήσατε τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης μέσω ατομικών ε, δικαιωμάτων ε, αλίας και είπατε ότι υπάρχει και ένα φάσμα ατομικών δικαιωμάτων, δεν είναι όλα ειδικιούς. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λογικά τα ατομικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων και των ITQ προσπίζονται από, τα, ε, από την αλληλεία υψηλού επίπεδου που έχει και μια δομή πολύ περισσότερο επιχειρηματική. Επομένως η δομή αυτή είναι πολύ πιο κατανοητή διότι μιλάμε για, με όρους οικονομικής απόδοσης, ε, δυνατότητας αλήψης κτλ. Αυτού οι μορφές τόλων είναι πιο κατανοητές και είναι πολύ πιο ευνοϊκές ε, για τη διαχείριση μέσω των ατομικών δικαιωμάτων. Διαπιστώνουμε όμως ότι υπάρχουν και αρκετές λήψεις για την ε, παράκτη αλληλεία και αρκετή δισταγμή αν θέλετε από πλευράς του τομέα της παράκτιας αλληλείας να δεχτούν αυτές τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να λειτουργούν και θα ήταν και το επιθυμητό. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς που γνωρίζετε καλύτερα το θέμα τι προσαρμογές ε, θα πρέπει να γίνει για ε, την ερασιτεχνική αλία, την παραδοσιακή αλία και την παράκτη αλία, ώστε να μπορέσουν να δεχτούν αυτό το σύστημα. Να προσαρμοστεί δηλαδή το σύστημα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να λάβει υπόψη ε, την παράκτη αλία και την παραδοσιακή αλία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό να δώσω το λόγο στους αγορητές για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους ετέθησαν. Θα ακολουθήσω την ίδια σειρά με τις παρεμβάσεις σας. Καταρχάς, λοιπόν, ο κύριος Βαλτιμάρσον από τη ΦΑΟ. Μπορείτε να απαντήσετε και να κάνετε όποιες παρατηρήσεις θεωρείτε ότι αρμόζουν στα όσα σας τέτοισαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω θα μπορέσω να απαντήσω σε ερωτήσεις Καταρχήν όσον αφορά τα ψάρια για ανθρώπινη κατανάλωση, όντως 44% ότι ο ψαριών αυτών προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο αριθμός αυτός βασίζεται ως επτοπλίστων ή στην τεράστια παραγωγή ή στην Κίνα και με, ε, προσφάτως έχουν μειωθεί οι αριθμοί αυτοί, αλλά είναι γύρω στο 45%. Όσον αφορά τα ηχθιάλευρα, υπάρχει μία σταθερή κατάσταση, δηλαδή το 1 τρίτο των αλλιευμάτων καταλήγουν σε ηχθιάλευρα και ε, ε, διάβασα για την ε, χρήση ηχθιαλεύρων στην υδατοκαλλιέργεια και από το 1996 έως το 2004 η χρήση των ηχθιαλεύρων για την υδατοκαλλιέργεια ήταν σταθερή. Άλλαξε το μείγμα διότι η τιμή ανέβηκε αλλά η κατανάλωση κατανάλωση έμεινε σταθερή και έχει υποκατασταθεί το ηχθιάλαυρο από άλλες ε, πηγές πρωτεϊνών όσον αφορά το σύστημα. Μιλώντας για την ε, ΦΑΟ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι η αφομοίωση των ε, δικαιωμάτων οφείλεται σε ορισμένες παραμέτρους Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να υπάρχει ιδιωτικοποίηση των αδειών αλληλείας και ποσοστός και μπορούν να τις ανακαλέσουν τα κράτη όπως η Ιρλανδία. Και ε, μια άλλη βασική παράμετρος είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα σύστημα αλλιευμάτων που θα δίνει μακροπρόθεσμα το δικαίωμα να αλλιεύει κανείς χωρίς όμως να είναι ιδιωτική ιδιοκτησία. Το δικαίωμα θα το διατηρεί το κράτος και θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να προσαρμοστείτε σε μια νέα περίοδο διότι δεν θέλετε να υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις στην αρχή και όταν πλησιάσετε στο τέλος των 10 ετών να μην ξέρετε τι θα γίνει παρακάτω. Βλέπω λοιπόν την κατάσταση όπως εμείς την ερμηνεύουμε και από ό,τι είπε και ο Χόιρουπ Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο χώρο. Αυτό όμως που είναι βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα και όσο πιο ισχυρά είναι τα δικαιώματα τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το σύστημα. Αλλά και υπάρχει και ένα πολιτικό ερώτημα. Αυτό επιθυμείτε. Εδώ θα τελειώσω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο ε, Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση που μου ετέθηκε αφορά κυρίως την παρακτιαλία. Στην παρουσίασή μου εγώ πρότεινα να γίνει μια διάκριση μεταξύ αυτού του οποίου παραδοσιακά αποκαλούμε παράκτη αλία η οποία διαφέρει από τη βιομηχανική αλληλεία. Και ε, θα πρέπει να το δούμε όχι από οικονομική σκοπιάς, αλλά να το εξετάσουμε με μια πιο κριτική ματιά σε αυτό το παλιό μοντέλο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εσωτερική αγορά και την ε, διάδοση των υποδομών επέτρεψε το νοπό ε, ψάρι το οποίο ψαρεύεται ε, στις παράκτης περιοχές να καταλήγει στην κοινή αγορά με τέτοια τιμή η οποία θα επιτρέπει στους πιο παραδοσιακούς αλείς να μην είναι οι παλιοί φτωχοί αλείς αλλά είναι πιο σύγχρονοι και να ευημερούν περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμώσουμε αυτή τη μορφή ανάπτυξης ε, στην παραδοσιακή παράκτη αλληλεία, την οποία εγώ αποκαλώ ε, αλληλεία πρώτης ποιότητας. Η αλληλεία είναι μια εμπορική δραστηριότητα η οποία επιτρέπει ε, την ε, προμήθεια των αγορών. Όμως η εμπειρία της Δανίας και η εμπειρία της Ισλανδίας αποδεικνύουν ότι εάν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ ε, αλλιευτικής δραστηριότητας και οικονομικής δραστηριότητας δημιουργούνται τεράστιες δυσκολίες διότι όταν υπάρχει πολύ ισχυρό οικονομικό συμφέρον αρχίζουμε να έχουμε παρεμβάσει στον τομέα από πλευράς ατόμων που διαβλέπουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα δικαιώματα αλληλείας ε, όταν ε, δε, δεν είναι και ιδιαίτερος ε, δαπανηρά και έτσι μονοπολούν τις δραστηριότητες. Και οι μικροί αλληλείς ε, έχουν περισσότερες δυσκολίες διαβίωσης, διότι Αυτή τη στιγμή ε, κάποιο μπορεί να ανακτήσει την εμπορική αξία του δικαιώματο αλλία που έχει αγοράσει, αυτό το δικαίωμα αλλία γίνεται ουσιαστικά μόνο ένα οικονομικό όφελο και δεν αντιστοιχεί πλέον σε κάποια δραστηριότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι νέες γενιές δεν έχουν δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας της αλίας. Το να θεωρείται συνεπώς το δικαίωμα αλληλείας ως ε, ε συνδεδεμένο σε ένα συγκεκριμένο είδο αποτελεί κίνδυνο για την παραδοσιακή και την παράκτη αλεία. Γι' αυτό ακριβώς και η συμβολή μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διάκριση σε δύο τομείς. Το τομέα της πιο περιφερειακής, ε, πιο παραδοσιακής αλίας που σχετίζεται με τον κλάδο και που επιτρέπει να γίνεται και μία κατανομή ποσοστώσεων, όχι ανασκάφος, αλλά να επιτρέπεται να γίνεται κατανομή σε ομοσπονδίες τοπικών αλλιέων, σε οργανώσεις τοπικών αλλιέων, ώστε ή αλληλεί σε κοινή συμμετοχή με άλλου να μπορούν να διαχειριστούν τις ποσοστώσεις. Στη Δανία έχουμε διαπιστώσει ότι το σύστημα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Και δεν πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο αντιβαίνει και στους κανόνες της αγοράς, διότι αυτές οι ποσοστώσεις ε, θα μπορούσαν να εκμισθώνονται και για κάποιο αντίτιμο ετησίως, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός στην αγορά. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια πιο φιλελεύθερη οικονομία σε σχέση με αυτήν η οποία ευνοεί το μονοπόλιο μεγάλων ε, ε, επιχειρηματιών που αγοράζουν όλες τις ποσοστώσεις τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν με το κεφάλαιο που διαθέτουν. Πρόταση δική μου λοιπόν είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μην κάνουμε αντιπαράθεση παραδοσιακής και βιομηχανικής αλίας, αλλά μετά βιομηχανικής αλίας και οικονομικά βιώσιμης, την οποία θα πρέπει να, στην οποία θα πρέπει να δοθεί μεγάλος αριθμός πόρων. Αυτός ε, κατ' εμέ είναι ένας τρόπος να προασπίσουμε τις τοπικές κοινωνίες και την ε, ε, παράκτια και παραδοσιακή αλληλεία με ένα καλύτερο όραμα προς το μέλλον. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ερώτηση που θα μπορούσα να απαντήσω εγώ. Αφορά τη συνέπεια τον τάξη στην ε, παράκτη αλία. Διότι η παράκτη αλής είναι σε δύσκολη θέση, αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια και ε, όσο υπάρχουν μεν επαρκείς ποσοστώσεις δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και οι παράκτη αλής δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να ε, κερδίσουν το ψωμί τους. Χρειάζονται μικρές μόνο ποσότητες. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τους κινδύνους ε, της κεφαλαιοποίησης των δικαιωμάτων αλληλείας μέσω της μεταφοράς τους. Θα ήθελα όμως να πω ότι αυτή είναι μία συζήτηση η οποία υπάρχει εδώ και πολύ καιρό διότι αυτή η κεφαλαιοποίηση οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές για τα πλοία. Κανένας αλλιέας δεν ε, αγοράζει ένα πλοίο εάν δεν έχει δικαιώματα και ποσοστώσεις. Ακόμη και στα κράτη-μέλη που δεν ε, αναγνωρίζουν αυτό τον τρόπο μεταβίβασης των δικαιωμάτων. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να το αποφύγουμε για ορισμένες δραστηριότητες και στο μέλλον και γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Τώρα, η μικρή αλληλεία αξίζει μια τέτοια προστασία. Νομίζουμε ναι, είναι ένα θέμα που μας επασχολεί εν πάση περιπτώσει, διότι μέσα στην ε, κοινοτική νομοθεσία τα μικρά πλοία αποτελούν 85% των πλοίων ε, και 9% μόνο 100 των αλλιευμάτων και 30% της αξίας. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να αποφύγουμε μία συγκέντρωση των δικαιωμάτων αλληλείας να επηρεάσει ε, στόλους που είναι σημαντικοί και πολιτιστικά και αλλιευτικά αλλά και από πλευράς ε, απασχολήσεως και προστιθεμένης αξίας. Νομίζω λοιπόν ότι η παρέμβαση του κυρίου Ρουτ τόνισε αυτή την πτυχή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν η αρχή είναι σωστή. Και μετά μπορούμε να βάλουμε και κάποιες επιφυλάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ε, Ευρωπαϊκής Αλίας ή διαφόρων περιφερειών ή τοπικών ε, αλληλευτικών κλάδων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χαούμπεκ που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αλλιών της Πολωνίας. Έχετε το λόγο για ένα τέταρτο, κύριε Ξέγκος Χαούμπεκ. Καλησπέρα σας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιώσω την ομιλία μου έχοντας υπόψη ότι μιλώ σε νεοεκλεγέντες ε, εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών, σε ένα νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε μια νεοπαγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε οι προτάσεις μας έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία γιατί τα προβλήματα που θα σας θίξω ήδη είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τις άμεσες επαφές που είχα όμως με τον ε, Επίτροπο Μπόρκ, δυστυχώς οι προτάσεις που υπέβαλα τότε δεν ε, ελήφθησαν υπόψη και τα προβλήματα μεταβιβάστηκαν, μετακυλίστηκαν στην ε, τωρινή κοινοβουλευτική θητεία και η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούνται τώρα με τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής μετά από τις, τους προσανατολισμούς της Πράσινης Βίβλου, έδωσα τον εξή τίτλο στην ομιλία μου. Η ανάγκη αλλαγών της, Ευρωπαϊ... της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση κάποιε κοινωνικέ και κοινωνικέ διαδικασίε μετά από την επιρροή υπερβολικής ε, νομικής ρύθμισης και έλλειψη διεξοδικών ε, επιστημονικών ε, μελετών στις λεκάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ κύριε Χαούμπεκ, επειδή διαβάζετε το κείμενό σας, να το διαβάσετε με λιγότερη ταχύτητα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσει κανείς ένα γραπτό κείμενο που διαβάζετε επιπλέον με μεγάλη ταχύτητα. Αν θέλετε λοιπόν να, να μεταφραστεί σωστά το κείμενό σας, παρακαλώ να το διαβάζετε λίγο πιο αργά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε πλήρω την αλληλευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στι αλληλευτικέ λεκάνε και του αλληλεί, είναι απαραίτητη μια προσεκτική ανάγνωση του εγγράφου που έχει τον τίτλο Ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, υπαριθμών 7 του 2007 για θέματα συστημάτων ελέγχου, επιθεώρησης και κυρώσεων σχετικά με την προστασία των κοινοτικών αλληλευτικών πόρων ε, μαζί με τις ε, απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω ότι αυτό το έγγραφο εκπονήθηκε σε ελεκτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται δηλαδή για ένα κοινοτικό έγγραφο. Το έγγραφο αυτό με ιδιαίτερα οξυδερκή και επαγγελματικό τρόπο περιγράφει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του ελέγχου σε έξι σημαντικά ελευτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα παρουσίασε μια σειρά ατασταλιών σε ό,τι αφορά την τήρηση του κοινοτικού ελευτικού δικαίου σε ορισμένες, ε, κράτες, ε, σε ορισμένες χώρες μέλη και μάλιστα ε, τέτοιε παρατυπίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο βαθιέ και σοβαρές που μερικές φορές είναι απίστευτο ότι συνέβησαν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να καταλάβει κανείς τις παρατυπίες που γίνονται στο κοινοτικό αλληλευτικό δίκαιο και μάλιστα είναι χαρακτηριστική μία παράγραφος από την τέταρτη σελίδα αυτού του εγγράφου αποτελεί εύγλωτη απόδειξη αυτών των ατασταλιών. Λέει λοιπόν αυτή η παράγραφος. Τα στοιχεία για τα αλλιεύματα δεν είναι ούτε πλήρη, ούτε αξιόπιστα, κάτι που παρεμποδίζει την εμπεριστατωμένη γνώση του Εύρου των αλλιευμάτων και ως εκ τούτου εμποδίζει και την σωστή εφαρμογή του συστήματος ε, των ΤΑΚ και των αλλιευτικών ποσοστώσεων. Ως εκ τούτου, το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι υποχρεωτικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη δεν εξασφαλίζουν ούτε την πληρότητα των ε, συγκεντρωμένων στοιχείων, ούτε αποκάλυψη των ασυνεπιών που υπάρχουν. Και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει με ε, ικανοποιητικό τρόπο των λαθών, τα λάθη και τις ανακρίβειες των στοιχείων των κρατών μελών, ούτε μπορεί έγκαιρα να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των αλληλευτικών αποθεμάτων. Σας επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ένα κοινοτικό έγγραφο που διευκολύνει και εμένα, γιατί μας ε, δίνει πολύ σημαντικές ε, προτάσεις για τα λάθη που υπάρχουν και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Τέτοιο λοιπόν ε, ε, πρόβλημα, όπως το επισημαίνει το ελεκτικό συνέδριο, δείχνει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σωστέ αποφάσει για την ελεκτική πολιτική, γιατί στερείται ακριβών και αξιόπιστων στοιχείων. Δεν γνωρίζει ούτε το εύρο των αλλιευμάτων, ούτε και τι διαστάσει των ε, αλλιευτικών πόρων. Οπότε, πώ να δώσει κάποιε προτάσει για μια διασφάλιση των αλλιευτικών πόρων. Οπότε ανακύπτει η ερώτηση, από τη στιγμή που μέχρι τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά είχε η ευρωπαϊκή αλληλευτική πολιτική, ήταν λογική τέτοια ριζική μείωση του αριθμού των αλληλευτικών σκαφών σε ορισμένε χώρε, μια και βάση για την πρόταση τη μείωση ήταν άγνωστη άγνωστη διάσταση των αλλιευμάτων καθώς και άγνωστες διαστάσεις των αλλιευτικών πόρων. Οπότε το έγγραφο αυτό που δεν περιλαμβάνει και τους ε, ελέγχους που γίνονται στη Βαλτική θάλασσα, δεν λέει τίποτα για την ε, λεκάνη της Βαλτικής. Παρ' όλα αυτά, αντίστοιχα νομικά προβλήματα υπάρχουν και στην περίπτωση της Βαλτικής, γιατί ανακριβείς ακριβώς στατιστικές πληροφορίες στρεβλώνουν την κατάσταση και την εικόνα για τα ελευτικά αποθέματα. Σημαντικά λοιπόν προβλήματα της αλίας είναι η υπερβολική νομοθετική ρυθμίση και συχνά αντιφατικές διατάξεις που είναι ακατανόητες και διαφορούν για τις βιολογικές ε, περιφερειακές και κοινωνικές ε, ιδιαιτερότητες των συνθηκών και μάλιστα γίνεται μία άνοθεν ε, προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης του ελευτικού δικαίου. Υπάρχει έλλειψη αντικειμενικών και περιστατωμένων επιστημονικών μελετών και ανακριβείς πληροφορίες και μάλιστα η ψευδικολογική προσέγγιση ορισμένων επιστημονικών κύκλων που χαρακτηρίζουν τους αλείς και την αλληλευτική προσπάθεια ως απειλή για το περιβάλλον. Η αδυναμία στις αντίδρασης επίσης ε, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των, οικολογικών, των ε, θαλάσσιων οικοσυστημάτων, κάτι που καθιστά αδύνατη μια ορθολογική αξιοποίηση του, των αλληλευτικών πόρων. Απόλυτη δυναμία ελέγχου στην, ε, στην αλία επίσης εκφυλισμός του αλληλευτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συνάφεια μεταξύ της νομικής θεωρητικής ε, ρύθμισης της αλίας αλλά και των ε, ε, συνθήκων που επικρατούν από οικονομική και βιολογική άποψη στις διάφορες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση συγκεκριμένων δικτύων για την αλίευση σολομού υπό το πρόσχημα και το επιχείρημα της μεγάλης θρησιμότητά τους για τις φώκενες. Ή η ανοχή και η υποστήριξη μάλιστα της αλίευσης ε, ε, για, για λόγους κτηνοτροφίας, για την Παρασκευή δηλαδή ε, αλεύρων κάτι που διαταράσει την βιολογική ισορροπία στην ε, λεκάνη της Βαλτικής. Δεν λαμβάνεται υπόψη σωστά οι προσδοκίες και οι ανάγκες των ε, περιφερειακών αλληλευτικών κλάδων. Ούτε δίνονται αποζημιώσεις σε περίπτωση περιορισμού των αλλιευμάτων. Γίνονται πολλές παρατυπίες και στις, περιβαλλοντικές, στις περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές και υπάρχουν πολλές παρατυπίες σε ό,τι αφορά την τήρηση του ελευτικού δικαίου, όπως δείχνει και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Όλες αυτές οι παρατυπίες που λαμβάνουν η χώρα στην Ευρωπαϊκή και στη Βαλτική, Αλία δείχνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Αλία. Βέβαια, είναι θετικό ότι ακόμη και ελεκτικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Αλία και ευελπιστώ ότι το ενεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντλήσουν τα κατάλληλα συμπεράσματα από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει αρκετή αποφασιστικότητα και αντικειμενικότητα για να αναζητήσει του υπέτειου τη σημερινή κατάσταση αλίας, όχι μεταξύ των Ευρωπαίων αλλιέων, αλλά ε, σε επίπεδο νομοθετικό. Γιατί η ποιότητα αυτού του, του, των νομοθετικών προτάσεων και η έλλειψη προσαρμογής τους στις περιφερειακές και βιολογικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την σωστή εφαρμογή τους στις διάφορες χώρες μέλη. Και μάλιστα ε, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, μιλούν κυρίως για την αλία χωρίς την, την Βαλτική θάλασσα, γιατί η Βαλτική θάλασσα συμπερίφθηκε στην κοινή αλληλευτική πολιτική μόλις την 1η Μαΐου του 2004, μετά την διεύρυνση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα προβλήματα των αλίων στη Βαλτική θάλασσα είναι ίσονος σημασία. Το αντίθετο, γιατί η ανεπαρκής γνώση των μεθόδων αλίας που επικρατούσαν πριν την διεύρυνση και η άκρητη υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά τη διεύρυνση επέτεινε τα προβλήματα στη Βαλτική. Μεταξύ των προβλημάτων είναι το πολύ σημαντικό πρόβλημα της αλίας για λόγου κτηνοτροφίας και παρασκευή ηχθιαλεύρων στη Βαλτική θάλασσα. Κάτι τέτοιο απειλεί την βιολογική και οικολογική ισορροπία ολόκληρης της Βαλτικής. Χρησιμοποιούνται σκάφη με ισχυρούς κινητήρες και μεγάλα δίκτυα με πολύ μικρά διάκαινα, μάτια, κάτι που οδηγεί σε υπεραλίευση μικρών διαστάσεων ε, ψαριών που είναι εκτός της ποσόστοσης. Παρά του, τα πολιτή προγράμματα διαφύλαξη των αληφτικών πόρων. Ασκείται δηλαδή μια αλία που ουσιαστικά είναι αντιαλία και αντιβαίνει πλήρως στο κοινοτικό δίκτυο δίκαιο και την προσπάθεια διαφύλαξη των αλληλευτικών πόρων. Όλα αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν τις νέες αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι όλα αυτά τα αλλιεύματα σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται. Γιατί κάποιοι πιθανοί έλεγχοι θα έδειχναν πόσο επιβλαβεί είναι αυτές οι δραστηριότητες και τι διαστάσεις έχουν. Κατά τη γνώμη των αλλιέων, αυτά τα αλλιεύματα για Παρασκευή χθιαλεύρων σε τόσο μικρή λεκάνη όπω είναι η Βαλτική είναι ανεπίτρεπτα, απαράδεκτα και θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως και να αντικατασταθούν από αλία πελαγικών ειδών μόνο για λόγους κατανάλωσης. Ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εισαγωγή της απαγόρευσης χρήσης των παρασυρώμενων απλαδιών για τον Σολομό με το επιχείρημα της θρησιμότητας που έχουν τα παρασυρώμενα απλάδια για τις φόκενες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν επιρροή αυτού του είδους των δικτυών ε, για τον πληθυσμό της Φόκενας. Ενώ σε άλλες σκανδιναβικές χώρες ε, ατιμόρυτα χρησιμοποιούνται τέτοια παρασυρώμενα πλάδια για την αλία Σολομού. Δεν υπάρχουν, παραλαμβάνω, ε, αποκαλυπτικά στοιχεία και μάλιστα στοιχεία του 2007 δεν έδειξαν ούτε ένα κρούσμα αλίευσης φώκενας σε παρασυρώμενα πλάδια για την αλία σολομού. Και παρόλα αυτά ισχύει η απαγόρευση χρήσης τέτοιων δικτών για το, δικτύων για το σολομό. Έτσι μειώθηκε και η ζήτηση άγριου σολομού σε ευρωπαϊκές ε, αγορές. Βλέπουμε κάποιες αλλοπρόσωλες μορφές και γελίες μορφές από την εφαρμογή του κανονισμού 1269 του 2009 που εγκρίθηκε και υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2009 από τον ίδιο τον Μανουέλ Μπαρόζο και που επιτρέπει να μην καταγράφεται η αλίευση γάδου γύρω από την Γκέτλαντ και μάλιστα δεν χρειάζεται κανείς να είναι ιδιαίτερα οξυδερκής για να αντιληφθεί ποιον συμφέρει και τι συμφέροντα εξυπηρετεί μια τέτοια πρόταση. Και είναι κρίμα που έγκυρα Ινστιτούτα όπως το ΣΕΦ επιτρέπουν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Και μάλιστα το μεγαλύτερο σκάνδαλο για τη διαχείριση της κοινοτική αλληλείας στη Βαλτική είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ε, αλλιεύματα από 6.000 περίπου σκάφη μικρότερα των 8 μέτρων δεν λαμβάνονται υπόψη στις ε, αλλιευτικές στατιστικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ε, ψαριού δεν συμπεριλαμβάνονται στα επιστημονικά στατιστικά στοιχεία. Κάτι που παραπεί τα στοιχεία και για την αλίευση αλλά και για την κατάσταση των αλιευτικών πόρων. Οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πεπισμένοι ότι οι κοινοτικέ θάλασσες και οι κοινοτικέ λεκάνες είναι ουσιαστικά βιολογικές έρημοι και απαιτούν κάποια προγράμματα ανανέωσης των αλληλευτικών πόρων που θα πρέπει να γίνουν φυσικά με κοινοτικά κονδύλια. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι όλες αυτές οι παρατυπίες κατά τη διαχείριση της κοινοτική αλίας οφείλονται στην άκρητη υιοθέτηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιστημονικού κεκτημένου τη Βαλτική Επιτροπή, του GBSFC το Ινστιτούτο αυτό με πολύ επιπόλο τρόπο έδινε επιστημονικές συμβουλές για την αλία πριν την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Και υπάρχουν πολλά έγγραφα που δείχνουν πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε, δεκτή αυτές τις, έκανε δεκτές αυτές τις επιβλαβείς ε, συστάσεις της ε, Επιτροπής της Βαλτικής που πολλοί επιπόλαιοι ελήφθησαν υπόψη για την αλία στη Βαλτική θάλασσα. Παρακαλώ, τελειώνετε, λέει η πρόεδρο. το document Έχω υποβάλει το έγγραφό μου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και δεν θα μπορέσω να το διαβάσω όλο. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία μεταρρύθμισης κοινής ελευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας πω κάτι που θλίβει ιδιαίτερα και πονάει τους Πολωνούς αλληλείς και που δείχνει κάποιες εσκεμμένες ενέργειες που γίνονται εις βάρος της Πολωνίας αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια αλόκοτη, ακατανόητη περίπτωση που κατά τη γνώμη των Πολωνών Αλλιέων είναι απίστευτη, ανεπίτρεπτη και πραγματικό σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα αυτό αφορά τη, τους ε, ελέγχους που γίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αλίας ε, με διακριτικό τρόπο εις βάρος των Πολωνών Αλίων. Να φανταστείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν στην Πολωνία 2.536 έλεγχοι σε αλληλευτικά σκάφη, ενώ ο αλληλευτικός ε, στόλος στη Βαλτική είναι ο μικρότερος στόλος, απαριθμεί μόνο 877 σκάφη. Ενώ ταυτόχρονα στην Σουηδία που έχει 1565 σκάφη στη Βαλτική, έγιναν μόνο 708 έλεγχοι και στη Φιλανδία που διαθέτει 3.196 ελευτικά σκάφη στη Βαλτική έγιναν μόνο 16 έλεγχοι. Μόνο 16. Τον ίδιο χρόνο, την τελευταία διετία. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ο έλεγχος αυτού του, ελέγχου, αυτού του οργανισμού ελέγχου ε, γίνεται και προγραμματίζεται από κάποιον. Ποιος είναι υπεύθυνο για την ε, υπερβολική αυτή επιθεώρηση που γίνεται στην Πολωνία. Γιατί γίνονται τόσοι έλεγχοι στην Πολωνία και όχι αντίστοιχοι έλεγχοι σε πολύ μεγαλύτερες αλληλευτικές δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως γίνεται παρενόχληση ορισμένων ε, μικροαλλιέων για να αποσπαστεί η προσοχή από τις πραγματικά μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλία που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες παρατυπίες. Είναι αποτελεσματικός ένας τέτοιος έλεγχος και αξιοποιεί με σωστό και ορθολογικό τρόπο τα κοινοτικά κονδύλια. Τις υπόλοιπες παρατηρήσεις μου μπορείτε να τις βρείτε στο εγγραφό μου που ήδη έχω υποβάλει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια το λόγο έχει η κυρία Κρίστχαν Στότυρ που είναι η σύμβουλος αλληλείας της ε, μόνιμης αντιπροσωπής της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι μπορεί να μας ε, παρουσιάσει ένα μοντέλο διαχείρισης, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Κρίστιαν Στότερ. Δυστυχώς εγώ καταλαβαίνω παλία, αλλά ονόματα σκανδιναβικών χωρών είναι πολύ δύσκολα για μένα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Γκούρι Κρίστιαν Στότυρ. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προφέρετε το όνομά μου. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ για να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το σύστημα διαχείρισης της αλίας της Ισλανδίας και πώς διαχειριζόμαστε εμείς τα θέματα της διατήρησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης του στόλου. Θέλουμε να σας δώσουμε μια εικόνα της ε, αλίας στην Ισλανδία στο πρώτο τμήμα και στο δεύτερο τμήμα ασχολούμαστε με τις πτυχές ε, του συστήματος διαχείρισης. Η χρήση των πόρων ε, στη θάλασσα γύρω από την Ισλανδία ήταν πάντα θεμελιώδους σημασία ε, για την οικονομική επιβίαση των Ισλανδών. Τα στοιχεία που έχετε εδώ καταδεικνύουν τα αλλιεύματα για τα βασικά είδη για το χρονικό διάστημα από το 1905 έως το 2007 η αλλιευτική βιομηχανία έφτασε στην ε, κορυφή της ε, στον 20ο αιώνα. Ξεκίνησε η μεγαλύτερη αλλιεύση στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και αυτή τη στιγμή αυξήθηκε ε, η αλληλεία ρέγκας και του προσφυγακίου το σύνολο των αλευμάτων της Ισλανδίας είναι γύρω στο 1,7 με 2,1 εκατομμύρια τόνους ετησίως και αντιστοιχούν στο 1,8 έως 2,5% των συνολιακών αλευμάτων παγκοσμίω. Περίπου 1.450.000 τόνους έχουμε ε, ετησίως και ε, πέρα από την ε, ζώνη επιτρεπόμενης αλήθειας της Ισλανδίας έχουμε περίπου 500.000 τόνους. Η ετήσια αξία της αγοράς των ε, αλευτικών προϊόντων, των θαλάσσιων προϊόντων, είναι γύρω στα 2 δις ε, δολάρια. Ε, αυτό το στοιχείο βέβαια δεν είναι ακριβές απόλυτα, διότι είχαμε και μια υποτίμηση της Ισλανδικής κορώνας. Να σας δώσω αυτό το διάγραμμα για να έχετε μια εικόνα ως προς το που βρισκόμαστε ως αλευτικό κράτος σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τα αλλιεύματα 15 ε, χωρών σε τόνους ε, και το συνολικό αλλιεύμα. Ε, η Ισλανδία ήταν το 2005 14η με 1,8 των συνολικών αλλιευμάτων παγκοσμίω. Η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο χωρών. η θαλάσσια ζωή και η χρήση της σε μεγάλο βαθμό έχουν δημιουργήσει την ποιότητα ζωής που απολαμβάνει η Ισλανδία σήμερα. Η αλληλεία είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα για την Ισλανδία από την ίδρυση της χώρας και για τον περασμένο αιώνα μπορούμε να δηλώσουμε ότι η ανάπτυξη της αλληλείας αποτελεί τη βάση της πρόοδου και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας παρά το γεγονός ότι η Ισλανδική οικονομία διαφοροποιείται συνεχώς, ε, εξακολουθεί να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλία. Εδώ έχετε ένα καταμερισμό της αξίας των προϊόντων ε, εξαγωγών της Ισλανδίας το 2007 ανατομέα αγοράς. Αυτό ε, αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η εξαγωγή αλλιευτικών προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι περίπου το 80% των συνολικών εξαγωγών. Όπως βλέπετε στο μικρό διάγραμμα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο σημαντική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο γάδος είναι το πιο σημαντικό είδος που εξάγεται. Ο Ασλανδικός στόλος αποτελείται από περίπου 103.000 ε, 103.000 ε, σκάφη ε, το μέγεθος του στόλου είναι περίπου σταθερό τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο στόλος της Ισλανδίας είναι πολύ ευέλικτος ε, ως προς τα ε, αλλιευτικά οργαλεία και επομένως είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε μια, έναν ακριβή καταμερισμό των σκαφών. Η Ισλανδία δεν επιβάλλει περιορισμούς ε, στο μέγεθος του στόλου. Ε, το ίδιο το σύστημα του ITQ αποτελεί κίνητρο για τους ε, παραγωγούς ώστε να προσαρμόζουν το στόλο τους ανάλογα με τις ανάγκες. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Δικαστήριο της Ισλανδίας έχει αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμό στον αριθμό ε, σκαφών. Κάθε σκάφος το οποίο πληρεί τις απαιτήσει αδειοδότησης ε, μπορεί να λάβει και μια άδεια λιλίας. Όταν ε, ελήφθη ο έλεγχος των 200 μιλίων το 1976, άρχισαν να υπάρχουν ανησυχίες ε, για υπεραλίευση των πιο πολύτιμων αλληλευτικών αποθεμάτων. Υπήρξαν, ε, υπήρξε εφαρμογή αρκετών περιορισμών και υπήρχε και μία έντονη πολιτική συζήτηση για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης έκτοτε. Το 1983 τα συστήματα ITQ τα οποία χρησιμοποιούνταν από το 1973 αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο το 1983 υιοθέτησε ένα ε, σύστημα διαχείρισης ατομικών μεταβιβάσεων ποσοστώσεων που βασίζονται στην απόδοση ε, αλίευσης τα, τα τρία τελευταία χρόνια και η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ήταν το 1984. Μέχρι όμως το 1990 υπήρχε μια επιλογή προσπάθειας ε, στο σύστημα που επέτρεπε να μειωθούν τα αλίευματα και να αξιολογούνται οι πόροι από το σύστημα ITQ το παρόν σύστημα, το οποίο είναι συνολικό σύστημα διαχείρισης, ακόμα βασίζεται στα ατομικά, στις ατομικά μεταβιβάσιμες ποσοστάσεις. Υπάρχει μία ε, νομοθεσία διαχείρισης για να δημιουργείται αποτελεσματική χρήση των θαλάσσιων πόρων και να επιτρέπεται η σταθερή εργασία και η βιωσιμότητα των ελευτικών κοινοτήτων. Στόχος λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε βιωσιμότητα των ε, αλλιευμάτων ενώ ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση στα οικονομικά ωφέλη του ελευτικού τομέα. Βάσει νομοθεσία, ε, τα μέγιστα επιτραπόμενα αλλιεύματα καθορίζονται από το Υπουργείο Αλλία και Γεωργία και η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη σύσταση του Θαλάσσιου Ινστιτούτου Ερευνών τα αλλιευτικά σκάφη λαμβάνουν ένα ε, σταθερό μερίδιο ποσόστησης ανάλογα με το ετήσιο επιτρεπόμενο αλίευμα. Και σήμερα ε, το 95% του συνολικού, της συνολικής αξίας των αλλιευμάτων περιλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα. Το Υπουργείο αποφασίζει ποια είδη ε, θα υπόκειται στο σύστημα του ITQ και όταν συμπεριλαμβάνονται και νέα είδη σε ένα σύστημα ατομικών μεταβιβάσεων ποσοστώσεων, υπάρχουν ε, ε, σκάφη τα οποία λαμβάνουν ένα μόνιμο μερίδιο ποσοστώσεων, το οποίο βασίζεται στα αλλιεύματά του των προηγούμενων τριών ετών. Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης της Ισλανδίας είναι η δυνατότητα μεταβίβασης. Η... Το μερίδιο ποσοστώσεων, που είναι το επίσημο ε, δικαίωμα ανάθεσης ποσοστώσεων μπορούν να μεταβιβαστούν ε, μέχρι 50% για κάθε αλλιευτική χρονιά. Και κάθε σκάφος ε, θα πρέπει να έχει μια άδεια αλλιεύσης εννοείται. Ε, οι ιδιοκτήτες που έχουν δικαίωμα αλληλείας πρέπει να καταβάλουν και κάποια αλλιευτική εισφορά και η συνολική εισφορά για κάθε χρόνο βασίζονται στα κέρδη του αλληλευτικού τομέα, καθώς επίσης και την ε, ανάθεση, την κατανομή των ε, αλληλευτικών αδειών. Ένας από τους τρεις βασικούς στόχους ε, του συστήματος διαχείρισης της Ισλανδίας είναι να διασφαλίσουμε ότι είναι αποτελεσματικός ο κλάδος, καθώς επίσης και ότι διατηρούνται τα θαλάσσια αποθέματα και υπάρχουν θέσεις εργασίας και βιωσιμότητα για όλη τη χώρα. Έχουν γίνει πολλές δυνατότητες εκλογήκευσης ε, και παγίωσης, αλλά υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες ότι κάποιοι χρήστες μπορεί να είναι πάρα πολύ, κάποιοι παραγωγοί μπορεί να είναι πολύ μεγάλοι και μπορεί να υπάρχει συγκέντρωση της αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο του 12% του μεριδίου των ποσοστώσεων που μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος παραγωγός ή κάποια, ε, κάποια οργάνωση αλλιέων. Και επίσης υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι τόνοι ε, ποσοστώσεων που κατανέμονται αναλόγως. Βασικός στόχος είναι να μην δημιουργείται ε, στρέβλωση στην αγορά και υπάρχει και ένα ειδικό προτιμησιακό καθεστώς ε, ε, για την αλληλεία με παραγαδιάρικα σκάφη που ευνοεί τους μικροαλίες. Η νομοθεσία απαγορεύει τις απορρίψεις και όλοι οι αλληλείς υποχρεούνται να εκφορτώνουν όλα τους τα αλλιεύματα. Ο βασικός κανόνας ότι όλα τα σκάφη είναι υποχρεωμένα να έχουν ποσοστώσεις αλλιεύσεως για όλα τα είδη και όλα τα, είδη, τα είδη υπόκειται στο σύστημα του ITQ και αν τα σκάφη δεν έχουν αρκετές ποσοστώσεις για τα αλλιεύματά τους, απαιτείται να τους ε, μεταβιβάζονται ποσοστώσεις από άλλα σκάφη. Αλλιώς μπορεί να ανασταλεί η άδειά τους. Υπάρχουν και κάποια ειδικά στοιχεία ευελιξία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο σύστημα ποσοστώσεων τη Ισλανδία. Όπω σα έχουμε ήδη δείξει, υπάρχουν μόνιμα μερίδια ποσοστώσεων τα οποία μπορούν να καταμεριστούν και να μεταβεβαστούν σε άλλα αλλιευτικά σκάφη. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ο κάθε αλλιέας να χρησιμοποιεί τα ετήσια ε, αιτήσει ποσοστό ποσοστώσεις ε, από ένα είδος και να τα αμοιβάζει σε άλλον και επίσης να κάνει και μια μεταφορά από ε, έτος αλληλείας σε έτος αλληλείας. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μέχρι το 33% στην επόμενη ε, χρονιά αλληλείας και μπορούν να υπερβούν τις ποσοστώσεις κατά 5%, ε, ποσοστό το οποίο στη συνέχεια μειώνεται από την κατανομή του μεριδίου τους της επόμενη χρονιάς πέρα από το σύστημα του ITQ που μαζί με την ε, κατανομή των πόρων αποτελεί το βασικό, τον ακροβωνιαίο λίθο της διαχείρισης του συστήματος, το σύστημα Θα συνεχίσω χωρίς διαφάνεια. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Χωρίς παρουσιάση, την παρουσίαση. Πέραν λοιπόν του συστήματος ITQ που μαζί με την ε, κατανομή των TAC ε, είναι ο ακρογωνιαίος λήθος του συστήματος αλλιεύσης, υποστηρίζεται και από διάφορα άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο κάποιων περιοχών, περιορισμός ε, σε αλευτικά εργαλεία και προστασία συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να διατηρούνται πολύ σημαντικοί βιότοποι. πέραν από τις επικρίσεις, ε, μάλλον συγγνώμη, μία από τις επικρίσεις του συστήματος ποσοστώσεων είναι το γεγονός ότι απορρίπτονται πολύ σημαντικά αλλιεύματα από τους αλληλείς όταν δεν έχουν ε, ιδιοκτησία σημαντικών ποσοστώσεων. Εδώ θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αναγνωρίζονται απορρίψεις σε όλα τα συστήματα διαχείρισης αλίας. Δεν βελτιώνεται το πρόβλημα και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η διαχείριση που βασίζεται στις ποσοστώσεις αλίες μας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες απορρίψεις ε, από ότι άλλα συστήματα. Η αλληλεία κατεστραμμένων ε, αλευμάτων ε, πολύ χαμηλής αξίας είναι δυστυχώς ε, παρενέργεια οποιασδήποτε μορφής αλίας και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να απορρίπτονται παρανόμως, ανεξάρτητα όμως από το νομοθετικό πλαίσιο, εάν δεν υπάρχει μια τιμή αγοράς που να τους επιτρέπει να τα πουλήσουν στην αγορά. Το θέμα αυτό ερευνάται στην Ισλανδία στον αλληλευτικό τομέα και πολλοί διοικητικοί φορείς αναζητούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να, μειωθεί αυτή, ε, να μειωθούν αυτές οι απορρίψεις που γίνονται για οικονομικούς λόγους. Αυτό οδήγησε στην ευελιξία της διαχείρισης, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, και υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι ε, τρόποι διαχείρισης περιοχών προκειμένου να προλαμβάνονται οι απορρίψεις. Οι αρχές της Ισλανδίας αναζητούν τρόπους για να εποπτεύουν και να μετρούν τις απορρίψεις ε, στην Αλία στην Ισλανδία. Αυτό θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για τη διαχείριση και ταυτόχρονα όμως και ιδιαίτερος δύσκολο. Από το 2001 το Ινστιτούτο Θαλασσών μαζί με τη Διεύθυνση Αλίας ε, κάνουν μετρήσεις για τις απορρίψεις στην Ισλανδική Αλία. Η συλλεγή δεδομένων στρέφεται κυρίως στην Αλία Γάδου και ε, κοκκινόψερ Νορβηγίας ε, και τα στοιχεία που έχουμε από το 2009 έως το 2007 καταδεικνύουν ότι οι απορρίψεις ήταν το 1,17% των εκφορτώσεων και αυτό για το γάδο και για το κοκκινόψαρο της Νορβηγίας είχαμε 3,82% των εκφορτώσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα της ατομικής μεταβίβασης ε, ποσοστώσεων έχει λειτουργήσει αρκετά καλά για να περιορίζουμε τα λιεύματα σε συγκεκριμένα όρια και θεωρούμε ότι το σύστημα λειτουργεί βάσει νομοθεσίας και όσοι ε, έχουν ενεργό ρόλο ε, στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται επίσης όρις είναι πολύ σημαντική η σωστή εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών και οποιαδήποτε αγαστή λειτουργία ενός συστήματος βασίζεται και στις εκφορτώσεις και στις μετρήσεις που έχουμε σε όλα τα λιμάνια της Ισλανδίας. Όταν έχει ζυγιστεί ένα λίευμα, από εκεί και πέρα καταγράφεται στην βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Αλληλείας και η βάση δεδομένων καταγράφει τη θέση αλλιευμάτων όλων των σκαφών στην Ισλανδία. Οι πληροφορίες είναι ανοιχτές ε, για όλους στο διαδίκτυο και αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαφάνειας και διασφαλίζει ότι γίνεται καλύτερος έλεγχος και εποπτεία της ε, θέσης των σκαφών ε, στην Ισλανδία. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το σύστημα ποσοστώσεων έχει λειτουργήσει καλά και μας επιτρέπει να ε, περιορίζουμε τα λιεύματα σε συγκεκριμένα όρια. Το σύστημα είναι ιδιαίτερο διάφανο, διότι με ελάχιστε εξαιρέσει ε, όλα τα αλλιεύματα εκφορτώνονται στην Ισλανδία και το 97% του συνόλου των αλλιευμάτων εξάγεται. Πριν συνοψίσω, θα ήθελα εν συντομία να σας πω κάποιες σκέψεις για τους βασικούς στόχους της πολιτικής αλλίας της Ισλανδίας, που είναι οι εξής. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμη χρήση όλων των θαλάσσιων πόρων, να κάνουμε κάθε δυνατό προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα των ωκεανών και των οικοσυστημάτων, να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αποφάσεις βασίζονται στις καλύτερες δυνατές επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες, να συμμετάσχουμε ενεργά σε διεθνή φόρα, να προάγουμε το ελεύθερο εμπόριο για τα ε, θαλασσινά προϊόντα και να διασφαλίσουμε ότι τα θαλασσινά προϊόντα της Ισλανδίας είναι ασφαλή και υγιεινά. Στην παρουσίασή μου σήμερα προσπάθησα να σας δώσω μια συνολική εικόνα της λειτουργίας ε, του συστήματος διαχείρισης της Ισλανδικής Αλληλείας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Νομίζω ότι για όλους είναι ενδιαφέρον μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας εξηγεί το σύστημα διαχείρισής της. Τέλος, πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, ο τελευταίος αγορετής είναι κάποιος ο οποίος είναι γνωστός σε όλους μας, ο κύριος Βίκμαν, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ την Europass. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φεύγετε. Υπάρχουν μέλη της Επιτροπής Αλίας που έχουν παραμείνει. Ε, αρκετοί, οπότε ευχαρίστως να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Έχω μία παρουσίαση η οποία σε λίγα λεπτά θα έρθει στην οθόνη, αν βέβαια λειτουργήσει η τεχνική, η τεχνολογία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσω στην ε, πολιτική European Organization for ε, representing the fishermen. Ε, στην πολιτική ε, ε, για τον στόλο και για τη διατήρηση εκπροσωπώ του, την Δανική Ένωση Αλλιέων και είμαι ο Γενικός Διευθυντής του οργάνου όπως επίσης και της οργανώσεως δανών παραγωγών αλλιέων και όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Σχετική Οργάνωση ε, είναι η ΑΚΦΑ και η APO συγκεντρώνει τους ε, αλληλείς παραγωγούς. Από όλες τις οργανώσεις Ε, έχουμε απαντήσει στην ακρόαση για την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρυσι και έχουμε όλοι ασχοληθεί στη Δανία με το θέμα αυτό και ε, υπήρξε μία απάντηση από την ΑΚΦΑ, από τις επιτροπές της, μία από την EAPO και επιπλέον εμείς έχουμε στείλει ε, από τα περιφερειακά συμβούλια απαντήσεις για λογαριασμό των κλαδικών οργανώσεων. Θα προσπαθήσω λοιπόν εδώ να παρουσιάσω ορισμένα σχόλια σχετικά με την πολιτική ε, στόλου και διατήρησης γιατί χρειαζόμαστε αλλαγή και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να ε, ακολουθήσει η ε, αλλαγή. Στην επάνω βλέπετε ε, ένα στόλο, αυτό δείχνει την ε, μείωση του στόλου. Βλέπουμε όμως ότι αυξάνονται τα αποθέματα και έχουμε το τζίρο ο οποίος ανεβοκατεβαίνει όπως συνήθως εις, ε, την, εις, εις βιομηχανίες τις βιομηχανίες τροφίμων. Ε, εξαρτώμαστε λοιπόν από τα τάξια και τις ποσοστώσεις που είναι οι κανονισμοί παραγωγής και επηρεάζουν πάρα πολύ τη Βόρειο Ευρώπη ενώ στην νότια πλευρά ε, της κοινή γεωληφτικής πολιτικής έχουμε μόνο περιορισμούς όσον αφορά την αλληλεία του τόνου. Οπότε δεν υπάρχει μία συνεκτική πολιτική ε, και ε, δεν χρησιμοποιούμε όλοι τα ίδια, ε, τις ίδιες μεθόδους. Επιπλέον πρέπει να δούμε πού μπορούμε να ψαρεύουμε, για πόσο χρόνο και όλα αυτά τα τεχνικά μέσα έχουν ε, ε, διευρυνθεί με τον αριθμό των ε, ημερών στη θάλασσα και των ορών, κιλοβατορών αλληλείας δηλαδή υπάρχει μία συνεκτική πολιτική διατηρήσεως των ειδών μέσω της αλληλευτικής πολιτικής και για να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, ε, τη στο δικό μου χώρο βλέπετε ότι οι αλλοίς ασχολούνται και στη Βόρειο Θάλασσα και περαιτέρω και ε, πέρα από το Σκάγερακ υπάρχει μια ειδική περιοχή. Νοτίως από εκεί είναι η περιοχή του Κάτεγκατ, επίσης συγκεκριμένη περιοχή. Μετά έχουμε την Δυτική Βαλτική και την Ανατολική Βαλτική και από πλευράς αλληλείας διαφοροποιούνται οι χώροι αυτοί όσον αφορά τους κανόνες, της πολιτικές διατήρησης αναλόγως των περιοχών και είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε διότι όταν μιλούν οι άλλοι ε, για την Βαλτική ασχολούνται, ε, αναφέρονται ιδίως στην Ανατολική Βαλτική και θα επανέλθω στο θέμα αυτό αργότερα. Επιπλέον ε, έχουμε την την ε, ε, αλία ε, όπου βλέπετε έναν κύκλο ο οποίος αποτελεί το σύνολο και έχουμε στην αρχή το ITQ για τα πελαγικά είδη και από την άλλη πλευρά έχουμε το ITQ για ε, ηχθιάλευρα και έλαια. Ε, μετά έχουμε ε, τον χώρο που υπάρχει η αλληλεία μόνο βάση αδειών, η μικρή αλληλεία και ε, υπάρχουν πολλά μικρά ψάρια ε, και όλα αυτά ολοκληρώνονται στην ε, βυθοπελαγική αλληλεία διότι πάντοτε όταν κάπου επεκτείνεστε κάποιος πρέπει να έχει κάποια μείωση και βλέπετε ότι αν υπάρχει κατανομή πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή αυτή. Έχουμε λοιπόν διάφορες ομάδες τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε αλλά κάποιος πρέπει να, τα, ε, ε, να πληρώσει τα σπασμένα. Οπότε ε, υπάρχουν πολλές συζητήσεις τις οποίες έχουμε σε εθνικό επίπεδο για να ε, σχεδιαγραφήσουμε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την πολιτική διατήρηση και ε, πόρων. Έχω μία επιστολή που μας έστειλε στις 5 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, αποδεικνύει αυτό που θέλω να εξηγήσω ότι ε, λέγουν ότι στην Δυτική Βαλτική πρέπει να πάψουμε να αλλιεύουμε τον Απρίλιο. Στην αρχή ε, θεωρούσαμε ότι ε, ο Μάιος που προβλέπτω στην αρχή δεν είναι σωστός ενώ ο, ε, ο Απρίλιος συνάδει με την εποχή αναπαραγωγής οπότε ε, είχαμε πει ότι αν είναι ε, παγωμένα ε, ε, στις θάλασσες το Φεβρουάριο και Μάρτιο γιατί δεν παίρνουμε μία ε, εξαίρεση για να πάμε στον Απρίλιο και μας είπαν όχι αυτό δεν είναι δυνατόν διότι είναι μία απόφαση του Συμβουλίου, ένας κανονισμός Συμβουλίου και πρέπει να σταματήσετε. Όπως σας είπα λοιπόν, ενώ κανονικά θέλουμε δύο ως τέσσερις μήνες για μία εξαίρεση, τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα χρειαστούμε δύο έως πέντε μήνες τουλάχιστον ε, επιπλέον αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να σας πω τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε από πλευράς πολιτικής και τώρα και στο παρελθόν. Δεν έχουμε ευελιξία ε, εάν ε, συμφωνούνται οι αποφάσεις ε, από πλευράς συν ε, αποφάσεως με το Κοινοβούλιο ή ε, κανονισμών από το Συμβούλιο. Και επιπλέον συζητήσαμε με τους δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου μας τι θα πρέπει να γίνει. Και ένας από αυτός ο οποίος αναφέρεται εδώ μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έχει δυνατότητα να λάβει αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα σε περιπτώσεις ε, έκτακτης ανάγκης. Λέει όμως ότι αυτό ισχύει μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν μιλάμε ε, για τα αποθέματα αλληλείας και όχι για τους αλληλείς. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία νοτέρα βία αν πρόκειται ε, για τα αλλιεύματα αλλά όχι για τους αλληλείς ε, και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην μελλοντική μας πολιτική. Ε, επανέρχομαι τώρα σε ένα θέμα το ε, οποίο ε, είναι η μεταφορά από τις ημέρες στη θάλασσα στην κατανάλωση ανά κιλοβατόρια διότι τα πλοία ή μάλλον οι χώρες σε πολλές κατηγορίες έχουν μία σειρά κιλοβατό ημέρων που μπορούν να αλλιεύουν και όταν αυτό θα ισχύσει παντού σημαίνει ότι ένα ε, μικρό αλλιευτικό από την περιοχή του Κάτεγκατ και Σκάτεγκατ είχε 158 μέρες αλλιείες το 2008 ε, και ε, μπορούσαν το 2009 να αυξήσουν κατά μία μέρα. Ε, με το σήμα όμως των κιλοβάτ θα μειωθούν από στις 180 σε 129 το 2010 και σε 113 το 2011. Υπάρχει δηλαδή μία αυτόματη μείωση 10% για την ανάκτηση των αποθεμάτων της Βορείας Θάλασσας. Υπάρχει μία μείωση και για το Κάτεγκατα αλλά και σε άλλες περιοχές. Παραδείγματος χάρη τις ακτές της Ιρλανδίας όπου βγάζουμε στο δρόμο τα πλοία αυτά διότι δεν μπορούν πλέον να ψαρέψουν τις ποσοστώσεις τις οποίες έχουν. Ε, το σύστημα είναι διαφορετικό στο Σκάγερα και στη Βόρειο Θάλασσα διότι εκεί θα μπορούν από 163 μέρες το 2009 να φτάσουν σε 67 μέρες το 2012 για να υπάρχει αποκατάσταση των αποθεμάτων. Δηλαδή ε, κλείνεται στους ανθρώπους αυτούς το μαγαζί τους ε, λόγω της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται. Έχω φέρει αυτό το διάγραμμα, ίσως δεν βλέπετε περί τίνος πρόκειται, αλλά είναι η τάση σε τον χωριοτικότητα από το 1992 στο 2009 των ε, κοινοτικών στόλων. Έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο, είχε καταρτιστεί τον Ιανουάριο, το παρουσιάσε η Επιτροπή το Φεβρουάριο σε μία συνεδρία που είχαμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ε, μείωση σε κιλοβατιμέρες ε, ε, που μπορείτε να ψαρέψετε εάν πάρετε τη δικιά μου χώρα όπου θα υπάρχει μία αύξηση ε, κατά 46% από το 90 ε, ε, για την Ισπανία είναι 40% για την Πορτογαλία 44% και καταλήγουμε έτσι σε μία κατάσταση όπου θα εφαρμόσουμε μία πολιτική η οποία είναι πολύ αρνητική για όλο τον τομέα διότι επιπλέον δεν μας επιτρέπει να έχουμε το χρόνο και καλές συνθήκες για τους εργαζομένους, δεν μας επιτρέπει να ψαρεύουμε ε, στα ανοιχτά παρά μόνο κοντά στις ακτές και πέραν αυτού για να σας ε, δώσω μία ενημερωμένη πληροφορία όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς θα πρέπει να ξέρετε ότι εδώ στην ε, Επιτροπή Αλληλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποια είναι η κατάσταση της αλληλείας σήμερα. Έχετε εδώ τρία διαγράμματα που δείχνουν το ποσοστό ε, για τον μπακαλιάρο, για ε, τον ε, αστακό και για τον πλάτακα και βλέπετε ότι η κρίση είναι πολύ σοβαρή ε, αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει μόνο να σκεφτόμαστε την πολιτική για την αποκατάσταση των αποθεμάτων και ε, για τους στόλους, αλλά να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και ευχαριστούμε κύριε Βίχμαν. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις προς το πάνελ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα διάφορα θα λάβουμε σύντομη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της για τα τεχνικά μέτρα. μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας ακρόασης περιμένουμε στα διάφορα την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μας παρουσιάσετε πολύ αποτελεσματικά ποιες ε, ε, δύσκολες καιρικέ συνθήκες υπάρχουν στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρειο Θάλασσα. Και ε, παρουσιάστηκαν και σχόλια από συναδέλφους σας ότι δεν είναι αλληλεία σε έναν κλειστό χώρο αλλά στη φύση και στις ακτές ε, όπου οι αλείς είναι εκτεθειμένοι στις ε, κακοκαιρίες. Επί μήνες λοιπόν μετά από τη διάσκεψη της Κοπεχάγης ξεκίνησε ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Η θερμοκρασία έπεσε απότομα και είναι ακόμη τα πάντα παγωμένα και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα λίευμα. Μετά λοιπόν αυτή την παγωμένη βελτιωμένη κατάσταση θα έρθει ο Απρίλιος και τον Απρίλιο, πολύ σωστά είπε ο κύριος Βίκμαν, θα υπάρξει ένας μήνας για την απαγόρευση του μπακαλιάρου και ε, του πλάτακα. Πράγμα το οποίο ε, μπορεί να ε, επηρεάσει το χώρο υπό διαφορετικές συνθήκες σε άλλες περιοχές. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν πολιτικά να δεχτούμε την ευρωπαϊκή πολιτική α, και να την ε, καταστήσουμε αποδεκτή στους αλληλείς μας. Γι' αυτό και κάνω μία έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το έγγραφο το οποίο έλαβαν οι αλληλείς από την Επιτροπή να το ξανασκεφτεί η Επιτροπή. Δηλαδή τι θα γίνει αν δεν μπορούν να δουλέψουν και να μπορέσουν να ψαρέψουν διότι πιστεύω ότι εφόσον η Βόρειο Θάλασσα είναι πολύ σημαντική για το χώρο μας αν δούμε την κατάσταση διαπιστώνουμε ότι εργαζόμενος χωριζόμαστε σε τρεις κατηγορίες και ότι η βόρειος θάλασσα είναι ε, ένα, μια περιοχή η οποία ουσιαστικά καλύπτεται από την παραγωγή της Βαλτικής και ε, υπάρχουν περιφερειακές επιτροπές οι οποίες έχουν δικαίωμα συναπόφασης αλλά θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για να γίνουν αποδεκτές. Τώρα έχουμε τον κύριο Ρομπάτσοκ. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Κρίστιαν Σδότηρ. Είπατε κυρία Κρίστιαν Σδότηρ ότι δεν χρειαζόμαστε τα ITQ και μετά μπλοκαρίστηκαν τα ITQ και μόνο 20% των ITQ χρησιμοποιούνται. Δηλαδή τι, κατάλαβα καλά, 80% των ITQ δεν χορηγούνται. Τι ακριβώς είπατε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και τι μορφή πιστεύετε θα έχουν, θα πρέπει να, τι μορφή θα πρέπει να λάβει στο μέλλον ο ελευτικός στόλος ε, στη Βαλτική θάλασσα. Thank you. Uh, I don't have any other speakers on my... Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. No. I'll still put another question. Εκτός αν παρέλειψα κάποιον, όχι. Και εγώ έχω μια ερώτηση προς την κυρία Κριστιαν Ντότερ. Είχα συνομιλίε πριν από λίγες εβδομάδες με πολιτικούς από τη νέα κυβέρνηση της Ισλανδίας και μου είπαν ότι θα εγκαταλείψουν το σύστημα των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων ούτως ή άλλως. Εκτός και δεν κατάλαβα καλά, μπορείτε να το σχολιάσετε. Βέβαια είναι πολιτικό αυτό το ζήτημα για την Ισλανδία και υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε. Σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις, Είπατε ότι το σύστημα των απορρίψεων λειτουργεί, δηλαδή δεν υπάρχουν πια απορρίψεις. Πώς όμως ε, ασκείτε την εποπτεία, την επιθεώρηση και είστε βέβαιοι ότι δεν απορρίπτονται αλλιεύματα από το στόλο. Τι κίνητρα δίνετε στα σκάφη προκειμένου να εκφορτώνουν όλο τους το αλλιεύμα γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο, να εξακριβωθεί ότι όντως δεν γίνονται απορρίψεις και όντως ε, όλο το αλίευμα εκφορτώνεται. Αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο μας προσκεκλημένο και μετά θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Προς τον Πολωνό συνάδελφο θέλω να πω ότι μόνο τα 200 πλοία από τα 1300 και της Φιλανδίας πια ασκούν δραστηριότητα. Ίσως γι' αυτό έγινε μόνο 16 έλεγχοι. Δεν έχουμε πια τόσο πολλά όσο αναφέρατε. Αυτό το σχόλιο προς τον Πολωνό συνάδελφο. Παρακαλώ απαντήστε στην ερώτηση του κυρίου Κούν και στις δικές μου αν έχετε την καλοσύνη. Mr. if you want to come. Κύριε Χαούμπεκ, θέλετε το λόγο για να σχολιάσετε και μετά να ακούσουμε τις απαντήσεις και των άλλων καλεσμένων. Εγώ προσπαθώ στις ομιλίες μου να απόσχω από προσωπικές ε, απόψεις και σχολιασμούς, ιδιαίτερα όταν έχω ε, κοινοτικά έγγραφα που δικαιολογούν τη θέση μου. Γι' αυτό μίλησα ε, για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα 1.356 φιλανδικά σκάφη, μόνο 16 έλεγχοι ασκήθηκαν σε φιλανδικά σκάφη την τελευταία διετία. Δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου όλα αυτά. Προτείνεται, μάλλον προκύπτει από, τις, από τα στοιχεία αυτά, μετά από τη διαίρεση 1356-16, ότι ένα φιλανδικό σκάφος ελιευτικό ή μία φυλαδική τράτα ελέγχεται μία φορά κάθε 400 χρόνια. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές και αυτή η διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε όλα τα κράτη που παραπονιούνται για ανεπαρκείς αλληλευτικές ποσοστώσεις. Αναφέρθηκε κάποιος ότι οι αλήσει έχουν μια φυσιολογική τάση να παρακάμπτουν το κοινοτικό δίκαιο. Εγώ θα σας έλεγα ότι ούτε τα κράτη, ούτε οι αλληλείς έχουν μια φυσική ροπή ε, παράκαμψης του κοινοτικού δικαίου. Αλλά μερικές φορές αναγκάζονται να το κάνουν. Και παρόλα αυτά, παρά την καράκαμψη, λειτουργεί η αλληλεία σε πολλές ε, αλληλευτικές λεκάνες, ξεκινώντας από τη Μεσόγειο και τε, καταλήγοντας στη Βαλτική. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση τι μορφή θα πρέπει να έχει η αλληλεία στη Βαλτική. Κάθε λεκάνη κάθε ελευτική λεκάνη, ανάλογα με το βάθος της, την ιδιαιτερότητά της, τα ελευτικά της είδη, τις κοινωνικές συνθήκες και τις παραδόσεις, θα πρέπει να τύχει ξεχωριστής μεταχείρισης, ιδιαίτερης. Πραγματικά μου σηκώνεται η τρίχα ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί μια ενιαία κοινοτική νομοθεσία για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Ξέρουμε ποια είναι τα ελαττώματα του εγγράφου που σας ανέφερα. Το επισημαίνει η ίδια ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ότι υπάρχουν παρατυπίες και ατασταλίε. Το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο επισημαίνει σφάλματα και ελαττώματα. Βέβαια, τα συμπεράσματα είναι τελείως αντίθετα. Ότι φταίνε οι αλληλείς και φταίνε οι χώρε. Νομίζω ότι μερικές φορές εξαναγκάζονται τα κράτη και αλληλείς να παρακάψουν το δίκαιο. Και μερικές φορές λειτουργεί ηλία ακριβώ επειδή δεν τηρεί το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι επιβιώνει. Σήμερα δεν είχα αρκετό χρόνο και έτσι δεν μπορούσα να αναπτύξω αυτό το επιχείρημα, αλλά νομίζω ότι έχω αποδείξεις για να στοιχειοθετήσω αυτό το επιχείρημα. Τώρα, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει η αλία στην Βαλτική. Είναι αρκετά ε, λεκάνη Στο 80% των αλλιευμάτων στη Βαλτική είναι ουσιαστικά γάδος. Και είναι και η ρηχή θάλασσα η Βαλτική. Μιλάω τώρα για το γάδο που πραγματικά εκφορτώνεται και όχι για τη θεωρία, για τα, για τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται για το γάδο στη Βαλτική. Άλλη θεωρία και άλλη πράξη. Επαναλαμβάνω, στη Βαλτική κυρίω ασκείται παράκτη αλία από μικρά σκάφη. Οπότε η αλία στη Βαλτική θα πρέπει να προσαρμόζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά αυτή τη ε, θαλάσσια λεκάνη, στα βιολογικά χαρακτηριστικά, στι δυνατότητε αναπαραγωγή συγκεκριμένων αλληλευτικών ειδών και στη συνεξάρτηση των αλληλευτικών ειδών. Οπότε στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η δυνατότητα βιομηχανικής αλληλείας στην Βαλτική με τεράστια δίκτυα βάθους άνω των 100 μέτρων, γιατί το μέσο βάθος της Βαλτικής είναι 60 μέτρα. Οπότε με τέτοια τεράστια δίκτυα, με κατακόρυφο βάθος 100 ε, μέτρα, ε, η αλία, η βιομηχανική που αλκείται σαρώνει τα πάντα. Αυτό δεν είναι αλία, αυτό είναι αντιαλία, αυτό είναι αντιοικολογία. Και αυτό γίνεται τελείως ανεξέλεκτα μερικές φορές. Υπάρχουν έλεγχοι για το τι συμβαίνει στα ελευτικά αυτά σκάφη. Δεν γίνονται καν έλεγχοι. Και μπορώ να σας αποδείξω αυτά που σας λέω. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δυνατότητε να προκαλέσει τέτοιου ελέγχου. Και αν έχει κάποιε αφιβολίε για αυτά που σα λέω, σα παρακαλώ να ζητήσει από το ελεκτικό συνέδριο να διενεργήσει συγκεκριμένο έλεγχο στη Βαλτική. Να ελεγχθούν όλε οι χώρε που αλλιεύουν στη Βαλτική. Γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν 1500 ελευτικά σκάφη και σαρώνουν τα αποθέματα ε, γάδου και δηλώνουν μόνο 325 σκάφη. Τα υπόλοιπα σκάφη τι κάνουν, τι αλλιεύουν. Ή έχουν δικαίωμα μόνο για 325. Δεν τα λέω αυτό για να σας σοκάρω. Δεν ε, έχω καμία σκανδαλοθυρική πρόθεση. Από τα ίδια τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις μελέτες προκύπτουν αυτά, τα ελαττώματα. Έχουμε τώρα νέο κοινοβούλιο, νέο, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει κατά, η κατάσταση να αλλάξει, να μην διονύσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Επίσης ε, είχαμε το σχέδιο ανάκαμψης των αλευτικών πόρων του Γάδου το 2007. Νομίζω ήταν άχρηστο αυτό το σχέδιο. Πολλά σφάλματα έγιναν στην αλληλευτική πολιτική. Θα πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε τη σελίδα. Πίσω μου κάθονται πολλοί Πολωνοί αλληλείς. Και αυτή την επίσκεψή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ως πρώτη επίσκεψη, ως την απαρχή διαβούλευσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες διαβούλευσης μας δίνει δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η αλία σε μια μικρή θάλασσα όπως είναι βαλτική θα πρέπει να είναι μικρή εμβέλειας. Δεν μπορεί να γίνεται βιομηχανική αλία για αλίευση ε, ψαριών για ηχθιάλευρα με τεράστια δίκτυα που σαρώνουν τα πάντα. Αυτό είναι αντιαλία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλιεύματα που ουσιαστικά συνιστούν αντιαλλευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χόλουμπεκ για την πολύ σαφή απάντησή σας και την εικόνα της Βαλτικής θάλασσας. Να περάσουμε τώρα στην κυρία Κρίσιαν Στόχτερ για να απαντήσει στις ερωτήσεις που της ετέθησαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για το ερώτημα για τους περιορισμούς για τη μεταβίβαση ποσοστώσεων. υπάρχει ένα μέγιστο μερίδιο ποσοστώσεων που μπορεί να είναι ιδιοκτησία ενός συγκεκριμένου αλιέα ή μιας οργάνωσης αλιέων. Μόνο το 50% το, ε, επίσης του επίσημου μεριδίου μπορεί να μεταβιβαστεί. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση για το κατά πόσον η Ισλανδία θα καταργήσει το σύστημα των ποσοστώσεων, Νομίζω ότι δεν τίθεται ούτε καν θέμα συζήτηση για την κατάργηση του συστήματο. Έχουν όμω υπάρξει κάποιε συζητήσει για ε, μια δεκαετή περίοδο ποσοστώσεων και όχι ένα ανοιχτό σύστημα όπω αυτό που έχουμε σήμερα. Και αυτό σχετίζεται και με τις συζητήσεις για το ε, τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των ποσοστώσεων, μάλλον που γινόταν πριν από 30-40 χρόνια όταν συστήθηκε το σύστημα. το Υπουργείο Λίας έχει συστήσει μια επιτροπή για να αναθεωρήσει το σύστημα και είναι όμως ακόμα πάρα πολύ νωρίς ε, για να κάνουμε εικασίες ε, κάνει για την ε, λειτουργία του συστήματος και τα αποτελέσματα της Επιτροπής. Όσον αφορά τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν για να διασφαλίσουμε ότι οι αλληλείς θα τηρούν τους κανόνες, πρώτον, οι αλληλείς υποχρεούνται να έχουν ποσοστώσεις για όλα τα είδη ε, τα οποία ε, εντάσσονται στο σύστημα ITQ και είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο έχουν στη διάθεσή τους για να προσαρμόσουν το καθεστώς των ποσοστώσεων μετά από την εκφόρτωση. Έχουν δηλαδή ένα ελάχιστο χρόνο για να αγοράσουν ποσοστάσεις ε, γύρω στις τρεις ημέρες μετά την εκφόρτωση. Επιπλέον, Υπάρχει μια διάταξη στην νομοθεσία που επιτρέπει να προσμετρώνται τα μικρά ψάρια μόνο για το 50% των ποσοστώσεων. Δεν έχω όλα τα στοιχεία τώρα μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα 5% του μεριδίου εντός ενός έτους αλίας ή κάτι αντίστοιχο. Και τρίτον, μπορεί να εκφορτωθεί ένα συγκεκριμένο ε, ποσό, ποσοστό χωρίς ε, ποσόστοση και να διατεθεί στην αγορά και το 20% των εσόδων πηγαίνουν μεν στον Αλιέα, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ε, οργανισμό ο οποίος έχει συσταθεί από το Υπουργείο και πάει για τις ερευνητικές μελέτες στη θάλασσα και μάλιστα ε, αυτό έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το, ερευνητικό ε, το Θαλάσσιο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ισλανδίας. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Και τέλος, ο κύριος Γουίκμαν δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει τις ερωτήσεις που του έγιναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τον Πολωνό συνάδελφο ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να επηρεάζει περισσότερο η κάθε περιοχή ε, της λήψη, τη λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να υπάρξει μία διαφορετική διάρθρωση λήψης αποφάσεων μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής Περιφερειών ο Γερμανός συνάδελφος αναφέρθηκε στις κακοκαιρίες στη Βαλτική. Όντως έχουν υπάρξει ε, διάφορα σοβαρά θέματα και νομίζω ότι θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι τα αποθέματα γάδου ε, εις την Βαλτική ε, εδώ και πολλά χρόνια δεν τα πάει καλά ε, και μειώνεται και αυτός είναι ο λόγος ε, γι' αυτό ζήτησαν να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης για να μην και δεν έχουμε ε, ας πούμε μειώσεις του χρόνου αλίες στην Ανατολική Βαλτική. Ο Πολωνός φίλος μας κατεφέρθη σκληρά στου τους κατά των αλλιέων και επειδή εγώ εκπροσωπώ όλους τους αλλιείς ε, εις ε, την Δανία ευχαρίστως σας έρθει στη χώρα μου να δει και τις, ε, τις συνθήκες και τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και τα διάφορα στοιχεία της οργανώσεως των αλλιέων της Βαλτικής όσον αφορά την κατάσταση με ε, τους πάγους. Μιλήσαμε και για τη διαχείριση των στόλων και ο Ισλανδός συνάδελφος δεν το ανέφερε, αλλά ίσως κάτι μας δίδαξε η Ισλανδία όσον αφορά α, τους στόλους, διότι δεν έχουν πολιτική στόλων. Αν έχετε ένα αλλιευτικό είναι πρόβλημά σας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό ή μεγάλο αλλιευτικό και θα έπρεπε να αφήσουν την αλληλεία την Ισλανδία με τα προβλήματά τους διότι εκεί υπάρχουν 200 μίλια χωρικών υδάτων ενώ στη Βαλτική και στη Σκανδιναβία είναι πολύ περίπλοκο το πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι πολύ ε, μεγάλο το έργο σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να την πολιτική πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 οπότε θα πρέπει να έχετε να μορφώσει όλα τα προγράμματα ανακάμψεως ε, και διαχειρίσεως θα πρέπει να έχετε αναμορφώσει τη βάση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, να έχετε αναπτύξει ε, νέους κανονισμούς για τα τεχνικά μέτρα, διότι προσπάθησε πέρυσι το φθινόπωρο να ξεκινήσει κάτι η Σουηδία, δεν τα κατάφερε ε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, άρα και αυτό εκρεμεί θα πρέπει να υπάρχει μία ε, νέα αναμόρφωση της κοινή οργανώσεως αγοράς. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα και το τέταρτο είναι ένας νέος κανονισμός ε, για το αλλιευτικό ταμείο, δηλαδή πώς θα πρέπει να αναμορφωθεί αυτό το διαρθρωτικό ταμείο. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο ένα-δύο επόμενα χρόνια, γιατί έχετε πολλά να κάνετε. Καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Βίχμαν. Σίγουρα θα χρειαστούμε τύχη. Αλλά οι πράσινες βίβλοι μας δίνουν πολύ κουράγιο και μας γεμίζουν με ενθουσιασμό. Τέλος, ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνω την ερώτηση. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι σχέση με αυτά που ακούσαμε κύριε Κουίφ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Να συγχαρώ καταρχήν τον Νίλ Βίχμαν που εντόπισε με πολύ εξωτερική τρόπο τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να τηρήσουμε τη δέσμη αυτή των κανονισμών που ανταποκρίνονται στα σχέδια και τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερη παρατήρηση αφορά τους ελέγχους. Εγώ ανήκω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ελέγχου του Βίγκο και ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κίνδυνο που έχει καταμετρηθεί. Οπότε, όταν ο πρόεδρος μιας ε, ένωσης αλλιέων ε, καλεί σε ανυπακοή του νόμου, <laughs> είναι λογικό να επιτείνονται οι έλεγχοι στη συγκεκριμένη αλία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να Υιοθετείται μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο νόμο και λιγότερες παρατυπίες ή διοικητικά τεχνάσματα για τα αλληλευτικά σκάφη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σοφή συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους Έλληνες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Quiff. And, uh, with the comment of the... ευχαριστούμε κύριε Κουίφ με τα σχόλια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα ήθελα εκ μέρου τη Επιτροπή Αλίας να ευχαριστήσω θερμότατα τους έξι καλεσμένους του πάνελ μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρουσιάσει και ομιλίε τους και είχαμε πολλές χρήσιμε συμβουλές γιατί αυτό ουσιαστικά χρειαζόμαστε. Και να σας ευχαριστήσω εγκάρδια και πάλι. Ολοκληρώνεται η δημόσια κρόση και θα περάσουμε σε λίγο στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Okay, members, we'll move on to, to any other business on... Ευχαριστώ. Να περάσουμε στα διάφορα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη και όπως είπαμε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να κάνει μια μικρή ανακοίνωση για την πρόταση που είχαμε το 2008 για τα τεχνικά μέτρα, η οποία κρεμεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Να δώσω λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Κουίφ από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε την ανακοίνωση. Η Γενική Διεύθυνση που εκπροσωπώ πρόκειται να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της για τα τεχνικά μέτρα που βρίσκεται επιτάπητος ε, από τον περασμένο Νοέμβριο στο Συμβούλιο ως συμβαστική πρόταση της Προεδρίας. Μία συμβαστική πρόταση που δυστυχώς δεν έγινε δεκτή εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της μετάβασης που έγινε από την παλιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περιλαμβάνει μία σειρά αρχών για τον τρόπο καλύτερης επιλογής των αλευτικών εργαλείων, της μείωσης των απορρίψεων και της προστασίας ε, του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τις συνέπειες ε, μιας υπερβολικής αλίας. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποσύρει την πρότασή της Κατά τη γνώμη μας, ε, μια τέτοια απόσυρση δικαιολογείται από δύο λόγους. Από τις διατάξεις της ηθίκη Λισαβόνας που επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το δικαίωμα πρωτοβουλία της να διαχωρίσει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη και άρα να μπορεί να εκχωρεί κάποιες αρμοδιότητες. Οπότε η πρόταση για τα τεχνικά μέτρα με τη μορφή που έχει σήμερα και όπως προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μετά την ε, γνωμοδότηση που έδωσε τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήγουν σε μία σύγχυση μεταξύ των ουσιοδών και των επουσιοδών στοιχείων. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να ανακαλέσει αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ουσιαδών από τα επουσιώδη στοιχεία όπω προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ένα δεύτερο λόγο που θα δικαιολογούσε την απόσυρση αυτή τη πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση για να κάνουμε μία ε, εις βάθος ε, εξέταση και των τεχνικών μέτρων δεδομένης της περιφερειοποίησης της κοινή ελευτικής πολιτικής για να εξακριβωθεί κατά πόσο αυτό το πλουστάσιο των εκτελεστικών μέτρων περιλαμβάνει μέτρα άμεση και αμεσης εφαρμογή και να γίνει μια σωστή διάκριση μεταξύ τους. Με την απόσταση αυτή δεν θα δημιουργηθεί κανένα κενό δικαίου. Γιατί το Νοέμβριο είχαμε αποφασίσει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να υιοθετήσει μεταβατικά μέτρα ώστε να εφαρμόζεται και με η τρέχουσα νομοθεσία και 18 μήνες μετά την ε, κατάργηση του κανονισμού 850 98. Οπότε, χάρη στα μεταβατικά μέτρα, θα συνεχιστεί η τρέχουσα νομοθεσία, εξασφαλίζοντας μια συνέχεια των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Και η μεταρρύθμιση αυτή, ανάλογα με το, με το πόσο θα διαρκέσει, δικαιολογεί, ίσως θα δικαιολογήσει αργότερα, ένα νέο αίτημα παράτασης ε, των μεταβατικών αυτομέτρων. Αυτό θα το δούμε εν καιρό. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Υπάρχουν άλλα σχόλια για την πρόταση αυτή της, Ευρωπαϊ... της ε, Γενικής Διεύθυνσης. Όχι, ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγγελία αυτής της πρότασης. Και περνάμε από τα διάφορα στις ανακοινώσεις ε, από τα συμπεράσματα της συνεδρίας των συντονιστών. Η Γενική Γραμματεία μας σας έχει υποβάλει τις προτάσεις των συντονιστών. Υπάρχει αίτημα των πρασίνων για μια μικρή αλλαγή στα πρακτικά. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο κατανομής των εκθέσεων. Οι πράσινοι θέλουν να αφαιρεθεί το τελευταίο τμήμα της φράσης που λέει θα πρέπει να κατανέμονται καταφθύνοντα τρόπο βάρους ή αριθμού μελών. Και αποφασίσαμε να στηρίζεται η κατανομή στα μόρια που διαθέτει κάθε ομάδα. Αυτό ήταν το αίτημα των Πρασίνων. Συμφωνείτε γιατί αυτή την αλλαγή των πρακτικών. Γιατί υπάρχει διαφορετική ερμηνεία στο ότι, στο συμφώνησαν οι συντονιστέ για το σημείο αυτό. Συμφωνείτε? Απλώς τροποποιείται η σειρά της κατανομή των εκθέσεων, τίποτα άλλο. Γιατί ούτως ή άλλως είχαμε συμφωνήσει για αυτό το σύστημα των μόριων των πόντων. Ωραία. Οπότε ε, γίνεται μια μικρή διόρθωση στα πρακτικά της συνεδρία των συντονιστών. Αυτά. Έχουμε και τις προτάσεις για τις επόμενες μα συνεδριάσεις. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.